Colleagues, please be seated. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Πολύ χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να κηρύξω την έναρξη των εργασιών μας αυτή τη δεύτερη μέρα της συνεδρίας μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη το εξετάζουμε από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και με την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οπότε καλωσορίζουμε εδώ τους Πρόεδρους και Αντιπρόεδρους. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντες πανελίστες εδώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κριστία για να μας εισαγάγει κάπως το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαστε στο σημείο 9 στην ε, ημερήσια διάταξη, έτσι, που πρόκειται για τη νέα στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και θα ακούσουμε τους εξέχοντες ομιλητές μας που είναι η κυρία Εντίτα Χέντρα πρώτα απ' όλα, που είναι Διευθύντρια για την Αμερική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Άντα Μουσούμπ, που είναι επιτετραμένος στην αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Στίβεν Πάιφερ, ο οποίος είναι ανώτερος εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Brookings. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι η παρουσίαση της νέας εθνικής στρατηγικής είναι πάντα κάτι πολύ σημαντικό για τις Προεδρίες των ΗΠΑ. Ξέρουμε ότι τέτοιες στρατηγικές δεν είναι πάντα σε επαφή με την πραγματικότητα. Απ' την άλλη είναι σαφές ότι αποτελούν ένα εργαλείο για το συντονισμό όλων των πολιτικών που είναι ζωτική σημασία εργαλεία. Είναι στρατηγική λοιπόν του Λευκού Οίκου μας ε, δίνει πολύ τροφή για σκέψη, ιδιαίτερα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς καμία αμφιβολία, πολύ χαιρόμαστε που επιβεβαιώνεται η διατλαντική σχέση στον τομέα κυρίως της ασφάλειας και της άμυνας. Επίσης χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε ότι γενικά η γλώσσα της στρατηγικής είναι πιο μετριοπαθής από ότι πολλά από αυτά που ακούμε στο δημόσιο χώρο. Επίσης, είναι κάτι που επιβεβαιώνει και διαφορές που υπάρχουν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαφανίζεται από τη στρατηγική το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα ενισχυτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η κλιματική αλλαγή δεν είναι και το μόνο στοιχείο κλειδί που λείπει από το έγγραφο αυτό. Υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα που λείπουν και η ανάμειξη της Ρωσίας στην εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν προσβλέπω από τη συζήτησή μας να ακούσουμε τους ομιλητές μας για το πώς βλέπουν τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μέλλον και να σχολιάσουν και την ανακοίνωση του Πρόεδρου Τραμπ για το ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιστρέψει στη Συμφωνία των Παρισιών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Άνταμ Σουμπ. Ο Άνταμ Σουμπ, πρώτα απ' όλα επιτετραμένος στην αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Οτίγκα, Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Έλερ, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας εδώ σήμερα και ευχαριστώ και τους άλλους προσκεκλημένους που ήρθαν επίσης. Χαίρομαι που ξαναρχόμαι εδώ και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική, έτσι όπως εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 2017, με υπότιτλο ε, κυρίως «Ρεαλισμός», βάζει προτεραιότητες, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ, πρώτα οι πολίτες μας. Αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν, είναι αντιμέτωπες μάλλον με έναν επικίνδυνο κόσμο και ότι πολλές εντάσεις ε, γίνονται όλο και πιο σημαντικές τα τελευταία χρόνια. Και στο συνδευτικό του γράμμα επαναλαμβάνει τις συντηρητικές αρχές, ε, στρατιωτικό κλάδο, οικονομία, ενίσχυση συνόρων, εμπορικές σχέσεις που βασίζονται σε δικαιοσύνη και αμοιβαιότητα. Συνεπώ, βεβαίω, και όσο κοιτάμε αυτή τη στρατηγική πρώτη Αμερική, γιατί μια τέτοια στρατηγική είναι, η Αμερική πρώτα, είναι το βασικό σύνθημα της νίκης της σημερινής κυβέρνησης, στόχο έχει να κοιτάει τον κόσμο με, ξεκάθαρα, ε, με ξεκάθαρο βλέμμα με νέα ματιά τους συμμάχους, τους εταίρους και στα σχόλια του για την ε, στρατηγική αυτή ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει ότι βρίσκεται αντιμέτωπη η Αμερική με έναν επικίνδυνο κόσμο, γιατί είναι ανταγωνιστικός, στρατικοποιημένος, οικονομικά επικίνδυνος και είναι κάτι το οποίο ξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Κίνα, Ρωσία αποτελούν πρόκληση για τι ΗΠΑ συχνά και μερικέ φορέ αναφέρεται ότι έχει αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων και μερικέ φορέ σε βάρο των Αμερικανικών συμφερόντων. Η στρατηγική λοιπόν απαντάει και λέει η Αμερική πρέπει να χρησιμοποιήσει ό,τι δυνάμει έχει, ενέργεια, στρατιωτικά, πληροφορίε κλπ. για να προστατεύσει του Αμερικανού, για να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα βάσει τεσσάρων πυλώνων. Ο πρώτος είναι εσωτερική προστασία, δεύτερον είναι ευημερία της Αμερικής, τρίτον είναι η ειρήνη και το τέταρτο είναι να ενισχυθεί η αμερικανική επιρροή. Σε μερικά αναφέρονται προτεραιότητες και δράσεις κατά τη διάρκεια του 2018, πρώτα απ' όλα προστασία των Αμερικανών. Αυτή είναι η βασική μας ευθύνη, να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς στην καθημερινή του ζωή. Οπότε κοιτάμε το θέμα της ασφάλειας στα σύνορα, αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών και μια ασφαλής Αμερική και όσον αφορά το κυβέρνο χώρο. Ο πυλώνος αυτός λέει ότι για να προστατευτούμε ε, σωματικά πρώτα απ' όλα και αναφέρεται αυτό και στα έγγραφα η Αμερική θα προσπαθήσει να προλάβει τις ε, απειλές προτού δηλαδή βρεθούν στο αμερικανικό έδαφος Επίσης αυξάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες, ασχολούμαστε με τον κυβέρνο χώρο και με την ε, άμυνα απέναντι στους πυράβλους αντιμετωπίζοντας όπλα μαζικής καταστροφής, με την καταστροφή τους και με ενίσχυση των δυνάμεων αντιμετώπισης τους. Μπορούμε να αναλάβουμε αμέσως δράση κατά τζιχαντιστών και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων για να μην υπάρχουν ε, συνωμοσίες, αντιμετωπίζονται τρομοκρατικά δίκτυα και γενικότερα τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι πρόθεση και ενίσχυση της αμερικανικής ευημερίας. Ο πρόεδρος λέει ότι η οικονομική ασφάλεια είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αναγνωρίζουμε ότι η δημιουργία μας βασίζεται στην εθνική μας δύναμη. Άρα πρέπει να είμαστε η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Θέλουμε διαφάνεια στην οικονομία, επίσης ανοιχτή οικονομία. Θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομία στη χώρα μας και να προσφέρουμε ένα ευνοϊκό διεθνές οικονομικό σύστημα που να συνεισφέρει στην ευημερία και την ειρήνη στον κόσμο. Και πρέπει να κάνουμε και περισσότερα με τους εταίρους μας στα διάφορα θεσμικά όργανα υπέρ ενός συστήματος το οποίο προστατεύει και βοηθάει να έχουμε ένα δίκαιο και ανοιχτό εμπόριο. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν μια οικονομική στρατηγική που θα ανανεώσει την οικονομία μας θα ενισχύσει τον Αμερικανό εργαζόμενο, θα ενισχύσει τις Αμερικανικές βιομηχανίες, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, καινοτομία, ε, τεχνολογικά προηγμένα επιτεύγματα, ελεύθερες ε, οικονομικές σχέσεις υπέρ της έρευνας, της καινοτομίας και θα προωθήσουμε την καινοτομία και όσον αφορά την εθνική ασφάλεια. Θα προωθήσουμε τις εξαγωγές των ΗΠΑ, θα ενισχύσουμε την καινοτομία, όπως είπαμε, θεμητός ανταγωνισμός και θα αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά. Επίση, αναφέρεται και το θέμα τη πνευματική ιδιοκτησία. Στην ενέργεια, επίση, θα προωθήσουμε τι εξαγωγέ μα για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μα, για ε, να προστατευτούμε από απειλέ. Επίσης, στηρίζουμε τη διαφοροποίηση στην ενέργεια, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην ίδια την Αμερική. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ειρήνη. Ο Πρόεδρος πιστεύει σε μια Αμερική ανανομένη που θα μπορέσει να διασφαλίσει περισσότερο ακόμα την ειρήνη. Η στρατηγική αυτή σημειώνει συγκεκριμένα την Κίνα και τη Ρωσία. Και χώρες όπως είναι η Βόρειος Κορέα και το Ιράν, χώρες Παρίες και γιατί λέει ότι εκεί υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες σχεδιάζουν επιθέσεις στην Αμερική και για να το αντιμετωπίσει αυτό η Αμερική θέλει να προωθήσει το ανταγωνιστικό της ε, πλεονέκτημα όσον αφορά την βιομηχανία. Αν υπάρξουν επιθέσεις στις ΗΠΑ θα τις αντιμετωπίσουμε και θα φροντίσουμε να μην μπορούν με βία ή με άλλο τρόπο να επιτεθούν στις ΗΠΑ. Θέλουμε επίσης ε, αποτρεπτική πυρηνική δύναμη. Όσον αφορά το διάστημα, θέλουμε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση για να στηρίξουμε τις ε, τηλεπικοινωνίες και τα οικονομικά δίκτυα με συστήματα πληροφοριών, με έλεγχο και περισσότερες δραστηριότητε από τον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε επίσης να απτύξουμε περισσότερο τι δυνατότητε μα στον κύβερνο χώρο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πληροφορίε που μα έρχονται από αντιπάλους μας που θέλουν να πλήξουν την ελεύθερη κοινωνία μας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε τις δραστηριότητε της Κίνας. Κοιτάμε επίσης τις ομάδες τζιχαντιστών και τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την κοινή γνώμη παντού στον κόσμο. Ε, ενισχύουμε και την διπλωματία μας. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, διπλωματικά, στρατηγικά μέσα, οικονομικά, ε, στρατιωτικά, όπως είπαμε, για να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας και να προστατεύσουμε τους συμμάχους μας. Το τέταρτο είναι ενίσχυση τη επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο. Μετά τον ψυχρό πόλεμο θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτού που αποζητούν την ελευθερία και την ευημερία, αυτού του λαού. Και είναι πολύ βασικό αυτό στι σχέσει μα και στου συμμάχους μα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προωθούμε την αμερικανική επιρροή στο εξωτερικό, λαμβάνοντα υπόψη την ευημερία και την ασφάλεια και με τους ε, συμμάχους μας, οι οποίοι έχουν μεγάλη σημασία για μας. Πρέπει με ελεύθερη βούληση να γίνονται σύμμαχοί μας. Σε αυτό το τέταρτο πυλόν θα ξεχρονίσουμε επίση τα οικονομικά μα μέσα, αμερικανικέ επιχειρήσει, ιδιωτικό τομέα, για να υπάρχουν νέε επενδυτικέ ευκαιρίε από άλλε χώρε. Θα χρησιμοποιήσουμε τη διπλωματία ώστε να επιλέξουν άλλε χώρε την κατάλληλη διακυβέρνηση κατά τη διαφθορά και υπέρ τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξουμε μεταρρυθμίσει υπέρ του ιδιωτικού κεφαλαίου και των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και υπέρ της προστασίας ε, των ε, λαών των χωρών αυτών. Θέλουμε να εμπνέουμε τους συμμάχους μας και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε ευάλωτες ε, χώρες και κοινωνίες. Δίνουμε προτεραιότητα σε ιδιαίτερα ευάλωτες χώρες όπως είναι το Αφγανιστάν για παράδειγμα. Θα δουλέψουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και σε πολυμερή φόρα με λογοδοσία, με βελτίωση των αποδόσεων στο ΑΕΜΕΦ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΠΟΕ θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αξίες που έχουμε στηρίξει μέχρι τώρα υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις κοινωνίες μας, με το κράτος δικαίου, με ενίσχυση των δικαιωμάτων της γυναίκας, στηρίζοντας τις μειονότητες και τα ατομικά δικαιώματα. Θέλουμε να δώσουμε ε, καλές εναλλακτικέ σε θρησκευτικές διανέξεις. Θα έπρεπε εδώ να αναφέρω ότι υπάρχει και μια παράλληλη στρατηγική που είναι η Εθνική Στρατηγική Άμυνας. Στις 19 Ιανουαρίου την ε, πήραμε αυτή από τον Υπουργό Άμυνας και λέει πώς θα... πώς θα φέρουμε την Αμερική περισσότερο σε κατάσταση εχμής και πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ανταγωνιστές μας. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερική πρώτα δεν σημαίνει η Αμερική μόνη της. Η στρατηγική δείχνει ότι μια από τη μεγάλη μας, μια μεγάλη μας δύναμη είναι ακριβώς η σύμμαχή μας, γιατί είναι κάτι το οποίο επεκτείνει ακριβώς την επιρροή μας και τη δύναμή μας. Μια ισχυρή και ελεύθερη Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Αμερική, για τη σταθερότητα και για την ευημερία εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Η Ευρώπη και η Αμερική έχουν ε, δεσμευτεί από κοινού υπέρ της δημοκρατίας, των ελευθεριών, των ατομικών και του κράτους δικαίου. Και φαίνεται από το άγραφα ότι θέλουμε να βαθύνουμε τη συνεργασία μας με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε ό,τι απειλές υπάρχουν στις κοινέ μας αξίες και αρχές και κοινή οπτική και κοινό όραμα. Αυτή είναι η στρατηγική λοιπόν που δείχνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να στηρίζουν την Ευρώπη, του συμμάχου μας, Και βέβαια περιμένουμε από τους συμμάχους μας στον ΝΑΤΟ να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, το δικό τους μερίδιο ευθύνης όλα αυτά. Η στρατηγική επαναλαμβάνει ότι οι συμμάχοι μας πρέπει να αυξήσουν στο 2% του ΑΕΠ τις αμυντικές τους δαπάνες. Τώρα για τη Ρωσία δύο λόγια ακόμα. Η Ρωσία αποτελεί μια μοναδική πρόκληση για μας και για τους συμμάχους μας και τέρους μας. Προσπαθεί να γίνει πιο ισχυρή, να επεκτείνει τα σύνορά της, υπονομεύει την ενότητα στο ΝΑΤΟ και προσπαθεί να παρέμβει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο ΝΑΤΟ. Προσπαθεί να εκφοβήσει τους γειτονές της με πυρηνικά, με τα ενεργειακά και με ανάπτυξη ακόμα περισσότερων στρατιωτικών ε, δυνάμεων. Κίνα τώρα. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με την Κίνα. Ξέρουμε βέβαια ότι θέλει στρατηγική θέση στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η Κίνα, που είναι μια ανησυχία για μας. Οπότε όσο πρατερότητα στις δράσεις μας, οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλει να συνεργαστεί με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία και τις απειλές που έχουμε από το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Η στρατηγική τονίζει επίση την αστάθεια που υπάρχει στη Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή, που έχει σαν αποτέλεσμα πρόσφυγε και μετανάστε για να αποφύγουν την αστάθεια και τον πόλεμο να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Εμεί ω ΗΠΑ βλέπουμε ότι δεν είναι ασφαλή η Μέση Ανατολή και κινδυνεύει ακόμα περισσότερο από του τζιχαντιστέ. Και θέλει μια σταθερή κατάσταση και σταθερή και ενεργειακή κατάσταση. Γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες για να ακολουθούμε τις σταθερές πρακτικές και με συνέπεια. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ε, ευρωπαϊκές επενδύσεις Μένες Πολιτής, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και αντιμετώπιση το θέμα του ανταγωνισμού και θέμα των πρακτικών από την Κίνα στην Ευρώπη. Αυτά περιμένει η Αμερική από την Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε πλήρη εφαρμογή του ελέγχου των ε, οπλισμών ώστε να έχει ουσία η προσπάθειά μας για έλεγχο των πυρηνικών. Συνεπώς, λίγα σχόλια ακόμα για το μέλλον. Ο Υπουργός Έλβεση ε, αναφέρθηκε τελευταία όσον αφορά το περιβάλλον. Ότι υπάρχουν ε, απειλές που επηρεάζουν ακόμα και την εθνική ασφάλεια. Ο Γκάρτνερ επίσης είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει απομονωτισμός. Όσο προχωράμε το 2018 θα δείτε τις δράσεις των ΗΠΑ, θα δείτε τον Ιούλιο στο ΝΑΤΟ θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το ΝΑΤΟ και τη συνεργασία μας εκεί και πλήρη εφαρμογή του ελέγχου των πυρηνικών όπλων. Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε για να έχουμε ενιαία προσέγγιση απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή από τον κόσμο που μπορεί να είναι απειλή για την ασφάλεια των κοινωνιών μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτά προ το παρόν. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και είμαι έτοιμο να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσει έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαμπ, για το γεγονός ότι μοιραστήκατε μαζί μας τις προτεραιότητες αμερικανικής πολιτικής και για το ότι μας παρουσιάσατε το έγγραφο για την Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ. Τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Εντίτα Χέρντα, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Διευθύνουσα Σύμβουλο για την Αμερικανική Ήπειρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, συνάδελφοι Άνταμ. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική στιγμή και για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα, έπειτα από τη δημοσίευση της στρατηγικής ασφαλείας και άμυνας της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε πού κατευθυνόμαστε και τι τελικά είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις διατλαντικές μας σχέσεις. Θέλω βεβαίως να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση της στρατηγικής σας. Ε, με διευκολύνατε, γιατί θα επικεντρωθώ στη δική μου ομιλία σε τρία θέματα. Πρώτον, πού βρισκόμαστε. Θα συγκρίνω την ευρωπαϊκή παγκόσμια στρατηγική με την αμερικανική αντίστοιχη και θα πω και κάποια λόγια για το ε, τι πιστεύουμε για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων. Ο Άνταμ βεβαίως ε, περιέγραψε πολύ σωστά την άνοδο της παγκόσμιας ε, τρομοκρατίας, την κατάσταση στη Συρία, τη μετανάστευση, ε, τη διέλευση των μεταναστών από τις ε, άλλες υπήρους, ε, την απειλή από κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ασφάλεια, υβριδικές απειλές, υβριδικός πόλεμος στην Ανατολική γειτονία, στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες που περιβάλλουν δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βεβαίως ε, ενισχύουν την επίγνωση που έχουμε ε, για την ανάγκη ενίσχυσης ε, της συνεργασίας Ένωσης και ΕΠΑ. Αντιμετωπίζουμε δύο επιλογές. Συγκρουσιακή λογική, αφενός, και αφετέρου τη σκληρή δουλειά που θα οδηγήσει σε αμοιβαία επωφελής λύσεις και πρέπει να διαλέξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαλέξει πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ισχυρός, αξιόπιστος εταίρος για εκείνους που θέλουν να υπάρχει μια επικοδομητική, ορθολογική συνεργασία στον κόσμο. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι μοναδική στο είδος της, καθώς ε, ε, περιλαμβάνει στρατιωτικές και μη στρατιωτικές πολιτικές. Όσον αφορά την Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις της για την Ευρω... ενωσιακή παγκόσμια στρατηγική, και πρέπει βεβαίως να, διαμορφώσουμε και εμείς τη στάση μας, πρέπει να πω ότι σε αδρές γραμμές η στρατηγική ασφαλείας ε, εξηγεί το τι σημαίνει το σύνθημα η Αμερική πρώτα. Όπως είπε ο Άνταμ, σημαίνει βεβαίως όχι μόνη της η Αμερική. Η... Το βασικό τμήμα, ε, το βασικό, ο βασικός στόχος της στρατηγικής ασφαλείας είναι βεβαίως η ανταγωνιστικότητα, η εμβάθυνση συνεργασιών και ε, η, ε, συντήρηση ε, τον, ε, και, ο σεβασμός στους ε, κανόνες που διέπουν το παγκόσμιο σύστημά μας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας θεωρούμε ότι έχει μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη όσον αφορά την ασφάλεια βεβαίως. Παρά το γεγονός ότι κά, κάποιες από τις διατυπώσεις στο έγγραφο για την Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας αντικοτοπτρίζει μεν κάποιες, κάποιες, κάποιους νεωτερισμούς και ε, γλωσσικές διατυπώσεις που θα επέλεγε ο Πρόεδρος, νομίζω ότι υπάρχει ταυτόχρονα μια συνέχεια με, με τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις. Αυτό που ε, θα πρέπει εμάς ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, μας απασχολεί είναι πώς θα εξασφαλιστεί ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε κανόνες και θα γίνονται σεβαστοί οι κανόνες αυτοί από όλους τους παίκτες και από την Κίνα και από τη Ρωσία. Και νομίζω ότι είναι μια θεμητή οπτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον κόσμο στον 21ο αιώνα. βεβαίω βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς συνεργασίας. Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλεία των ΗΠΑ ε, διατυπώνει το στόχο ε, να τεθεί επικεφαλής η Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής, ε, και την ενίσχυση της ε, οικονομικής της ευημερίας ως εργαλείο για την εξασφάλιση της ασφάλειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Και ε, σε αντίθεση με την αμερικανική πολιτική, η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας δίνει περισσότερη έμφαση στην κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εύρυθμη λειτουργία της ε, ε, δημοκρατίας, αντίθεση με την Αμερική, αμερικανική στρατηγική, η οποία δίνει περισσότερη έμφαση στην, ε, στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές ανάμεσα στις δύο στρατηγικές. Ωστόσο, αυτές οι, διαφορε... διαφορές στρατηγική δεν πρέπει να αναιρέσουν την καλή συνεργασία, τις ε, κοινέ ευκαιρίες ε, και τις κοινέ αξίες που έχουμε στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η ίδια η, ιδέα του ρεαλισμού βάσει αρχών, μια από τις ε, βασικές σκέψεις και έννοιες που εισάγει αυτή η νέα στρατηγική, τον είπα, αναφέρει ακριβώς αυτόν τον ρεαλισμό ε, στην, ε, στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Επανεπιβεβαιώνει ότι ε, η αμερικανική πολιτική δεν εγκαταλείπει βασικές αρχές τις οποίες έχει ακολουθήσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Εσωτερική ανθεκτικότητα αυτό είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στην, εθνική, στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Στην αμερικανική στρατηγική ε, αναφέρεται ο ίδιος ο όρος, ωστόσο αφορά βεβαίως μόνο την, ε, τη χώρα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάντως υπάρχουν ε, αναφορές ε, προσήλωσης στους διεθνείς οικονομικούς φορείς, Συμφωνία Bretton Woods και αναφέρεται και η ανάγκη μεταρρύθμισης των ε, διεθνών φόρα. Και εδώ βεβαίως υπάρχει κοινό έδαφος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θεσμικά όργανα και οι διεθνείς οργανισμοί βεβαίως κατά την αμερικανική αντίληψη ε, θεωρούνται ως ε, φόρα ανταγωνισμού για το ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή. Για την... Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας αναγνωρίζει την, την ανάδειξη νέων απειλών, όπως είναι οι υβριδικές απειλές, η κυβερνοασφάλεια. Η δε κυβερνοασφάλεια τονίζεται ως κρίσιμης σημασίας ε, ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση με τις πυρηνικές κεφαλές ε, σήμερα είναι πιο ε, περίπλοκη από ό,τι στον ψυχρό, ψυχρό πόλεμο. Χρειάζεται, αναφέρεται στη στρατηγική, ε, ενίσχυση και αξιοποίηση της διπλωματίας και άλλων ε, οδών πολιτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν από οι ρωσικές προσπάθειες αποδυνάμωσης της διατλαντικής συνεργασίας. Η οικονομία λοιπόν θεωρείται ως βασικό στοιχείο για την ασφάλεια, την καινοτομία και την ε, έρευνα. Σε αυτό συμφωνούμε και εμείς. Εκεί άλλωστε αναφέρεται και στη δική μας ε, παγκόσμια στρατηγική η ευμερία ως εργαλείο για την, εξασφάλιση, για την προστασία της ασφάλειας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έννοια του ρεαλισμού βάσει αρχών και αυτός κατά την εθνική στρατηγική ασφαλείας και κατά την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας είναι ε, ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε στην από εδώ και πέρα συνεργασία μας. Τι θα γίνει από εδώ. Η διατλαντική συνεργασία και οι σχέσεις βεβαίως εξακολουθούν να είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε στρατηγική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, ισχυρός και αξιόπιστος πάροχος ασφαλείας στο διεθνές σκηνικό και βεβαίως ε, έχει σεβαστεί ε, και την ήπια δύναμη, τη μη στρατιωτική δύναμη, τον είπα, ε, στην ανοικοδόμηση χωρών. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, Χρειάζεται μια, ε, μια συνεργασία, μια συμμαχία στον τομέα της ασφαλείας και της άμυνας και έργο που θα επιτρέψει στα κράτη μας να αξιοποιήσουν καλύτερα τον προϋπολογισμό άμυνάς τους και την αναγνώριση βεβαίως και τη συμβολής που έχει Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ως εταίρος της ε, Εθνικής στρατηγική Άμυνας των ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες, αποτελεί δείγμα για όλα αυτά. Η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ ΕΕ, είναι βεβαίως απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι του 21ου αιώνα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε, μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Ε, Παρ' όλα αυτά τα θεμέλια της διατλαντικής συνεργασίας παραμένουν στιβαρά και νομίζω ότι ο εκπρόσωπος, ε, τον, η ύπατη εκπρόσωπος μάλλον, ε, το δήλωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η διατλαντική συνεργασία έχει βαθιές ρίζες και η φιλία μεταξύ των ευρωπαϊκών και του αμερικανικού λαού είναι πολύ ισχυρή και υπερβαίνει τα όρια των κυβερνήσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δεν μπορούμε ούτε να ε, αντιδράσουμε υπερβολικά σε περιστασιακές ή και πρόσκαιρες αλλαγές στην πολιτική των, ΗΠΑ όταν γνωρίζουμε ότι οι βασικές αρχές που διέπουν αυτή την πολιτική παραμένουν αμετάβλητες. Ευχαριστώ πολύ. Για αυτά που είπατε. Κρατάω το πρώτο Αμερική, αλλά όχι η μόνη της. Και τώρα έχω την τιμή να δώσω το λόγο στον κύριο Στίβεν Φάιφερ από το Brookings, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, εξόχοντα μέλη της Ευρωβουλής. Με χαρά βρίσκομαι σε αυτό το πάνω σήμερα να συζητήσουμε τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την ασφάλεια. Είμαι στο Brookings ως πανεπιστημιακός, αλλά να σας πω ότι δεν μιλάω εξ του Brookings, αλλά είναι προσωπικές οι απόψεις μου. Θα κάνω καταρχά τέσσερι γενικέ παρατηρήσει για την εθνική στρατηγική ασφάλεια και μετά θα κάνω συγκεκριμένα σχόλια για το πώ ακριβώ αυτή η στρατηγική αφορά την Ευρώπη και ιδιαίτερα Η γενική αυτή στρατηγική νομίζω περιλαμβάνει μια γενική άποψη των απειλών που αντιμετωπίζουν η ΕΠΑ, όπω επίση, και το πώ θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι απειλέ. Αντανακλά μια κύρια ρεπουμπλικανική κομματική προσέγγιση αυτή η πολιτική. Και βέβαια αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί συντάχθηκε από το στρατηγό Μακμάστερ, το Γενικό Σύμβολο Ασφαλεία, και δεν αποτελεί έκπληξη τη στιγμή που ο αντιπρόσωπο έχει συγκεκριμένε πολιτικέ απόψει από αυτού, ο κ. επίση, ο Υπουργό Άμυνα κτλ. Δηλαδή το έγγραφο αυτό ξεκάθαρα κάνει μνήα στο πρώτο Αμερική, στο America First, αλλά βεβαίως είναι αυτονόητο αυτό τη στιγμή που είναι ένα έγγραφο εθνική ασφαλείας. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι η εθνική πολιτική ασφάλεια, όχι μόνο αυτή, αλλά όλε γενικότερα, σκεγγραφούν την προσέγγιση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση κυρίων πολιτικών και προκλήσεων ασφάλεια. Γενικά περιλαμβάνουν μια κάτωψη, μάλλον με παγκόσμια άποψη και περιγράφουν το πώ θα μπορούσαμε να θα το μετωπίσουμε όλα αυτά. Καταρχά, έχουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για την πιθανή αμερικανική πολιτική σε κάποια σενάρια. Εγώ ήμουν 27 χρόνια ως σε διάφορες θέσεις ως Αμερικανός διπλωμάτης, ασχολήθηκα με διάφορα θέματα που αφορούν πυρηνικά πρόθεση ας πούμε, της οικονομικής πολιτικής στην Ουκρανία, επικοδομικές σχέσεις γειτονίες με το ΝΑΤΟ στη Ρωσία κτλ. Και όταν είχαμε αυτές τις πολιτικές, πάντοτε εντάσσονταν στη γενικότερη στρατηγική εθνική ασφαλείας. Δεύτερη παρατήρηση για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν μου είναι ξεκάθαρο ότι άμεσα συμφωνεί με κάποια στοιχεία κλειδί αυτή τη προσέγγιση εθνική πολιτική ασφαλεία. Παραδείγματο χάρη και θα αναφερθώ λεπτομερέστερα σε αυτό στη συνέχεια. Η Εθνική Στρατηγική ασφαλεία ε, παρουσιάζει μια εικόνα τη ε, ε, Ρωσία που εμφανίζεται ω αντίπαλο των ΗΠΑ και τη Δύση. Είναι σωστή αυτή η εκτίμηση κατά την απόψή μου, Όμω, η περιγραφή στην Εθνική Πολιτική ασφάλεια και οι συστάσεις για την Αμερικανική απάντηση και όντω η προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει η ΗΠΑ σε σχέση με την Ρωσία τα τελευταία χρόνια μου φαίνονται αρκετά διαφορετικές από τις απόψεις του Προέδρου που έχει εκφράσει μέχρι τώρα και όταν έχει αναφερθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς δεν είμαι, κατά το... δεν είμαι κατά πόσο το έγγραφο αυτό παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα για τις προθέσεις του Προέδρου σε συγκεκριμένα σενάρια που πρόεδρος που ακολουθεί, μπορεί να ακολουθήσει μια πιο εξειδικευμένη πολιτική και απαντήσεις και ανταποκρίσεις πέρα από αυτό που λέει δημοσίως στα tweet. Έχουμε λοιπόν ένα στοιχείο προβλεψιμότητας, κάτι το μη προβλέψιμο και αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι και θετικό. Νομίζω ότι πραγματικά εξυπηρετείται καλύτερα η Αμερική όταν οι δράσει είναι προβλέψιμε. Στι περισσότερε περιπτώσει, οι ΗΠΑ θέλουν φίλου οι φίλοι μάλλον και οι ενδεχόμενοι εχθροί να καταλάβουν το τι προτίθεται να κάνουν οι Αμερικανοί και τι όχι. Αυτό αφορά τους φίλους και τους συμμάχους μας, αλλά είναι κρίσιμο βεβαίως και για τους πιθανούς αντιπάλους, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ε, αποτροπή συγκεκριμένων καταστροφικών δράσεων εκ μέρους των αντιπάλων. Έχουμε λοιπόν αυτή την, αυτό τον αυξανόμενο οικονομικό, στρατιωτικό και βιομηχανικό ανταγωνισμό και κυρίως έχουμε τις προκλήσεις που θέτουν η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρειος Κορέα και το Ιράν. Και βεβαίως ε, εδώ περιλαμβάνεται και το γεγονό ότι αυτές οι χώρες ε, είναι ανθεωρητικές σε σχέση με την παγκοσμία τάξη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας τη συμβολή των ΗΠΑ στην δυτική ασφάλεια ε, κάτι το οποίο αφορά την καθηγητική τάξη ε, μέσω των ε, οργανισμών ή θεσμών όπως το ΝΑΤΟ, διάφορες άλλες υπηρεσίες, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί και οι θεσμοί, έστω και αν είναι ατελείς και παρουσιάζουν αδυναμίες, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη τα τελευταία 70 χρόνια. Και η διατήρηση αυτών των θεσμών πράγματι και η ενίσχυσή τους πράγματι μου φαίνεται ένας, αδμε... ένας ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης προκλήσεων που προέρχονται από Κίνα και Ρωσία ενδεχομένω. Η Εθνική λοιπόν Στρατηγική Ασφάλειας δεν το υπογραμμίζει αυτό το σημείο και μάλιστα φάνηκε ότι αυτό ήταν ε, μια πρόθεση εκ των συντακτών να προσαρμοστούν στις απόψεις του Προέδρου, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ συμμαχίων και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών για τη ΣΥΠΑ. Τώρα να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια για το πώς ακριβώς ε, εμπλέκεται εδώ η Ευρώπη σε σχέση με αυτές τις προκλήσεις, ιδιαίτερα σχέση με τη Ρωσία. Και θα συμφωνήσω ότι αυτή η εθνική στρατηγική ασφαλείας καταρχάς ε, λέει ότι μια ελεύθερη και ισχυρή Ευρώπη είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ. Έχουμε το άρθρο 5 της ε, Ιδρικής Συμφωνίας του ΝΑΤΟ όπου τονίζει κυρίως ε, τα θέματα ασφάλειας και άμυνα σε σχέση με το ανατολικό κομμάτι. Έχουμε την Ρωσία, η οποία προσπαθεί να ασκήσει επιρροή, προσπαθεί να προσπάσει ε, φίλους και εταίρους από τη, τον από την Ευρώπη και να ξεσθενεί στο ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα έχουμε την αύξηση του στρατηγικού δυναμικού τη Ρωσία, έχουμε τον εξυγχρονισμό των ε, πυρηνικών δυνάμεων στρατηγικών και μη στρατηγικών της Ρωσίας και ε, έχουμε και προσπάθεια της ε, Ρωσία να παρενέβει στι εσωτερικέ πολιτικέ δημοκρατικών χωρών. Περιγράφει αυτό το έγγραφο επίση και μια Ρωσία η οποία ανταγωνίζεται την Δύση και προσπαθεί να αντιστρέψει την παγκόσμια τάξη μετά την εποχή του, του ψυχρού πολέμου. Η εθνική λοιπόν στρατηγική όταν προσιάστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ προλάβανε και την ενίσχυση των σχέσεων και τη συνεργασίας με την Ρωσία. Αλλά αυτοί που παρακολουθούν τις σχέσεις της Ρωσίας, είπα, θα ήθελαν πραγματικά να δουν μια ουσιώδη συνεργασία μεταξύ των δύο. Όμως είναι δύσκολο αυτό να γίνει χωρίς να υπάρξει αλλαγή στις ε, προβληματικές συμπεριφορές του Κρεμλίνου που οδήγησαν στο χαμηλότερο σημείο των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης ε, μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και νομίζω αυτό ε, το είπαν αρμόδιοι όταν είπαν ότι εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη στάση της Ρωσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιθετική της στάση σε σχέση με την Ουκρανία. Η Αμερικανική απάντηση τώρα ετοιμότητα, στρατιωτική, εξεχρονισμό των πυρηνικών και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ξέρουμε επίσης ότι το Πεντάγωνο βέβαια θα αντιμετωπίσει δημοσιονομικούς περιορισμούς για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μετά η στρατηγική μιλάει για την σημασία της αναβάθμισης των αμερικανικών διπλωματικών δυνατοτήτων παγκοσμίω και αυτό είναι ένας από του λόγου για του οποίου υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αίσθηση αδράνειας και αδυναμίας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να περιλάβουμε εδώ και τις δράσεις κατά του ξεπλήματος και άλλων δράσεων και νομίζω ότι επ' αυτή η ελληνική πολιτική έχει ενισχυθεί προσπαθώντας δηλαδή να τονίσουμε ότι αν υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τις κυρώσεις προς τη Ρωσία αυτές θα πρέπει να δεθούν από άλλα μέτρα. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και με τις ε, κυβερνοεπιθέσεις, παρόλο που θα ήθελα να αναφερθώ και σε άλλα σενάρια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, είπα, να αναζητήσουν τρόπους αποτροπής της επιρροής της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο ε, μετά από αυτά που έγιναν το 2016. Εγώ ανησυχώ τώρα το Κρεμλίνο και μετά από αυτά που έγιναν το 2016, νομίζω ότι τα κατά είναι περισσότερα από τα υπέρ και δεν ξέρω κατά πόσο θα το επαναλάβουν. Τώρα με μονομένες βέβαια δράσεις έχουν κάποια λογική, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι ένα είδος έλλειψης στην εθνική στρατηγική. Δεν αφορά μόνο τη Ρωσία, αλλά και άλλες περιοχές. Η στρατηγική μιλά για το πώς ακριβώς οι ΙΠΑ θα έπρεπε να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Όμως δεν περιγράφει ένα γενικότερο πλαίσιο Αντιμετώπιση τη ε, Ρωσία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρωσία, αλλά γενικά με αυτή η στρατηγική μιλά για τη Βόρεια Κορέα και τι προκλήσεις που παρουσιάζει η Βόρεια Κορέα. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο, διαβάζοντας το εγγραφό, κατά πόσο η αμερικανική ανταπόκριση ή απάντηση θα ήταν η αποτροπή, οι διαπραγματεύσει για τη μείωση του πυρηνικού δυναμικού ή, ή κάποια σύγκρουση για την ε, καταστροφή αυτού του δυναμικού. Πρέπει λοιπόν αυτές οι προσεγγίσεις για τη Ρωσία να περιλαμβάνουν την αποτροπή και τη στρατιωτική αλλά και στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να πιέσουμε σε καταστάσει όπως η Ουκρανία αλλά και τρίτον θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα συνεργασία με την Ρωσία όταν υπάρχει σύγκληση συμφερόντων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Βεβαίω. Είναι πολύ σημαντική η κοινή προσέγγιση με την Ευρώπη. Αυτή η συνεργασία όχι μόνο είναι απαραίτητη, αλλά ενισχύει και την Αμερικανική διπλωματία και την Ινδική διπλωματία γενικότερα. Δηλαδή, η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΕΕ τα τελευταία χρόνια για τι κυρώσει στη Ρωσία ήταν πολύ σημαντική μετά από την ρωσική επίθεση κατά τη Ουκρανία. Έστειλε ένα μήνυμα στήριξη, αλλά και δυτική αλληλεγγύη. Και παρόλο που αυτά τα μέτρα, αυτέ οι κυρώσει δεν έχουν αποτρέψει το Κρεμλίνο από την οπτική τη τάση του στην Ουκρανία, νομίζω ότι έχουν μελλοντική αποτροπή για περαιτέρω ενδεχόμενε ε, δράσεις στο μέλλον. Επίσης, να πω ότι αυτή η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας έχει βεβαίω κάποιε, ελλείψει, αλλά οι κύριε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΙΠΑ στη Δύση ε, περιλαμβάνονται. Έχουμε στρατηγική, αλλά ξαναλέω δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο αυτή η στρατηγική προβλέπει την ανταπόκριση, την απάντηση ή τη στάση του Προέδρου Τραμπ σε συγκεκριμένε περιόδους κρίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέσβη Σαμπ Πάιθερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ανοιχτές σας παρουσιάσει για τόσα μας είπατε όσον αφορά την εθνική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε και στη στρατηγική εθνικής ε, άμυνας. Κατά πάσα πιθανότητα ε, θα μπει στο πρόγραμμά μας κάποια στιγμή και θα ασχοληθούμε και με αυτήν. Είμαστε κάπως αργοί, αλλά πάση περιπτώσει μας ενδιαφέρει. Τώρα, συζήτηση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Έλερ, μια που είναι ο πρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας μας ε, για τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τόσο νωρίς το πρωί και μόνο με ένα καπουτσίνο τι να σας πω, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά θέλω να μας θυμίσω λίγο, ακούγοντας και τα επίμαχα ζητήματα, το Αν καθίσετε με τους Ρώσους και με τους Κινέζους και ακούσετε τη δικιά τους εθνική στρατηγική, και υπάρχουν και εκπρόσωποι από τα think tanks, οι απόψεις θα δείτε ότι δίστανται. Νομίζω, από τη δικιά μου την πλευρά τουλάχιστον, ότι η δημοκρατική τάξη που πρέπει να δημιουργήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Και θέλω να επιθυμίσω λίγο, πέρα από τα συνήθη πολιτικά, και κάτι ακόμα. Η εθνική στρατηγική από την ε, στρατιωτική οπτική γωνία δεν είναι κάτι καινούριο. τα προβλήματα παραμένουν και επικεντρωνόμαστε εξίσου σε αυτά. Καμία ευρωπαϊκή χώρα ή η ευρωπαικη Ένωση δεν θα μπορούσε να αναπτύξει στρατιωτικές ε, λειτουργίες ε, εξίσου χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση κατά του Ατλαντικού. Όμως κατά την άποψή μου αυτό που είναι αρκετά ανησυχητικό είναι ακριβώς ότι δεν γίνεται μνήα στην Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή δεν κάνει τη σύνδεση με το γεγονός ότι όταν ε, η Ευρώπη, η και είναι σταθερή, ε, τότε και οι Ηνωμένε Πολιτείε ευημερούν και είναι σταθερέ. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Παρόλα αυτά δεν αναφέρεται στη στρατηγική η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα και αναφέρεται μόνο ως απειλή για τη Ρωσία, που είναι μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία βέβαια για το πώς βλέπει κανείς την Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια. Οπότε κατά τη γνώμη μου λείπει και αυτό το συμβολικό στοιχείο στα πλαίσια των πολυμερών πολιτικών γιατί αλλιώς αποδυναμώνονται και ο ΠΟΕ και τα Ηνωμένα Έθνη. Στον ΠΟΕ η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντιπροσωπεία, μιλήσαμε με το Κογκρέσο, ε, συζητήσαμε με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και το ρωτήσαμε ξανά και ξανά και τα μέλη του Κογκρέσου ποια θα είναι η αμερικανική πολιτική για να ορίσει νέα μέλη στο δικαστήριο του ΠΟΕ, που είναι πολύ βασικό για το σύστημα. Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με τις Ηνωμένε Πολιτείε, παρόλο που εκείνος υποστήριξε ότι είναι πιο πολύ θέμα διαδικασίας. Αλλά εμείς λέμε ότι επηρεάζει την κατάσταση απ' άκρη σ' άκρη, μέχρι την Κορέα. Γιατί είναι πράγματα που θα επιλύσουν διενέξεις που θα προκύψουν τον 21ο αιώνα δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική, έχει να κάνει με την ασφάλεια, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη άλλων περιοχών στον κόσμο για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες λύνουν τα προβλήματα σε ένα πολυμερές σε πλαίσιο, αλλά ειρηνικά. Και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Οπότε η ερώτησή μου είναι εξή. Όλα είναι έτσι transactional. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τους δικαστές, βλέπει το θέμα των δικαστών ε, στον ΠΟΕ, έτσι τότε όλα τίθενται σε αμφισβήτηση. Θα ήθελα λοιπόν κάποια αντίδραση και είναι μια διένεξη που πάει πολύ πιο βαθιά από ό,τι νομίζουμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Έλμαρ που είναι εισηγητής της, ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Όταν λέτε ότι η Αμερική πρώτα, πρώτα η Αμερική δεν σημαίνει μόνη η Αμερική, βεβαίως είναι αλήθεια. Διότι γνωρίζετε όμως, γνωρίζετε όμως ότι αν όλοι πούμε η χώρα μου πρώτα, τότε όλοι μόνοι μας θα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μια λογική αντίφαση λοιπόν σε αυτό που είπατε. Και ο επιτετραμένος ε, που μας παρουσίασε τα τέσσερα σημεία, αν τα εξετάσετε ένα προς ένα, αφορούν όλα το αμερικανικό εθνικό συμφέρον. Πουθενά δεν αναφέρεται η ε, δεν αναφέρονται οι πολυμερείς σχέσεις, ε, οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού και επίσης δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει και μια σημαντική διάσταση της ε, σύγχρονης ασφάλειας. Ξέρουμε ότι η ασφάλεια δεν αφορά μόνο τα στρατιωτικά ζητήματα στο σύγχρονο κόσμο. Αφορά το κλίμα, το περιβάλλον, το εμπόριο, και τι αντίστοιχε πολιτικές. Και εδώ, ε, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν τεράστιες αντιφάσεις. Α εξετάσουμε το θέμα της Αφρικής, για παράδειγμα. Αν δεν αναγνωρίσουμε την κλιματική αλλαγή και υπάρξει ερημοποίηση περαιτέρω περιοχών γύρω από τη Σαχάρα, αυτό θα επηρεάσει και ε, την πολιτική ασφαλείας και την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας. Το, το TPP για παράδειγμα δεν αφορούσε μόνο από την άλλη μεριά το εμπόριο ή το περιβάλλον. Ε, επρόκειτο για μια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών του ειρηνικού ένας, ένα, ένα, μια, ένα πλαίσιο δηλαδή φιλίας για όλες αυτές τις χώρες. Η αποχώρηση λοιπόν από τις σχετικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ δημιούργησε ένα τεράστιο κενό. Κάτι που με τη σειρά του θέτει κίνδυνο και την ασφάλεια. Και επίσης αναβαθμίζει και το ρόλο του Πεκίνου ως προς την προστασία της ασφάλειας στον ειρηνικό χωρίς βεβαίως να το επιδιώκει μια τέτοια στάση, είναι όμως παράπλευρη απώλεια και αυτό. Και εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές καλούμαστε να ε, ε, να πάρουμε θέση στον πόλεμο και στον ανταγωνισμό που διεξάγεται ανάμεσα στο Πεκίνο, τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον. Στην ε, Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ αναφέρεται ρητός ότι οι σύμμαχοι της, ε, των ΗΠΑ πρέπει να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ στις παγκόσμιες προσπάθειες τους. Πουθενά όμως δεν γίνεται λόγος ε, για κοινέ προσπάθειες στη βάση κοινών συμφερόντων. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχω πολύ σημαντικές αμφιβολίες όταν αναιρούνται δηλαδή αρχές στις, των διαθλαντικών σχέσεων που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον ότι ο βασικός υπερασπιστής της ε, ασφάλειας εξακολουθεί να είναι για εμάς το ΝΑΤΟ, όμως είμαστε σε θέση, αν το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιτελέσει πλέον αυτόν τον λόγο, να πάρουμε και δικές μας πρωτοβουλίες. Η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρος. Εντάξει, εγώ είχα λίγο παραπάνω καφέ από το συνάδελφο τον κύριο Έλλερ. Άκουσα τα σχόλια και νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό το οποίο ήδη είπατε, τη διαφορά δηλαδή ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. Και η σημασία που έχει του να είναι κανείς αξόπιστος και προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή σκηνή. Τα λόγια με τις πράξεις διαφέρουν πράγματι. Έτσι καλλιώς τα λόγια δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παίκτη στη διεθνή σκηνή. Όμως, τι είναι τα λόγια, πολύ συχνά είναι τα περίφημα tweets. Υπάρχει όλο αυτό το έγγραφο του NSS, της Εθνικής Στρατηγικής, και μετά έχουμε τα tweets τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα οι Ηνωμένε Πολιτείε να γίνονται ένας μη προβλέψιμος παίκτη. Δεύτερον, το θέμα των κανόνων στους οποίους βασίζεται η διεθνής τάξη, που είναι πολύ βασική. Γιατί πολιτικά υπάρχει κατακαιρματισμός ανά τον κόσμο. Αν μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτούς τους κανόνες που εξελίσσονται μεν, αλλά πάση περιπτώσει είναι καθορισμένοι για το πώς οργανώνεται η διεθνής ε, τάξη. Αν κάποιος υπονομεύει τους κανόνες αυτούς, αυτό προμηνεί πολύ κακούς καιρούς. Χρειάζεται η καλή μορφή, ναι, αλλά χρειάζεται και στήριξή τους και όχι υπονόμευσή τους. και αυτά που είπατε για το Υπουργείο Εξωτερικών που δεν καταφέρνει να κάνει αυτά που πρέπει. Και η δράση και αντίδραση με χώρες ανά τον κόσμο είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Και έχω τώρα δύο πράγματα για δύο χώρες. Αναφερθήκατε στο Αφγανιστάν. Πέρυσι είδαμε το υψηλότερο επίπεδο δυσκολιών, σοβαρή επιδείνωση όσον αφορά το Αφγανιστάν. Και υπάρχει και το GCPA που με φέρνει πίσω στην αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα. Ιράν, δηλαδή, και συμφωνία για τα πυρηνικά. Όλοι ασχολούμαστε με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιρροή του Ιράν στις γύρω χώρες. Συμφωνία, τι σημαίνει. Σημαίνει κάνουμε μια συμφωνία, εμένουμε σε αυτήν και φροντίζουμε όλοι να την κάνουμε να λειτουργήσει αυτή η συμφωνία και όχι ξαφνικά έτσι από μόνοι μας ε, φεύγουμε. Γυρνάμε την πλάτη σε αυτήν. Ευχαριστώ. Συντονιστέ τώρα. Ο κύριος Γκάλερ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Έλα μόλις το είπε. Δεν υπάρχουν πολλά καινούρια ουσιώδη σημεία στην στρατηγική ασφαλείας. Τουλάχιστον όμως χαιρόμαστε που επαναλαμβάνετε την προσήλωσή σας στο ΝΑΤΟ. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό το ότι χρειάζεται και να το πούμε. Ε, από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια ολόκληρη άλλη διάσταση η οποία επίσης πρέπει να επισημαθεί. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΠΕΣΚΟ έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ε, και το χρέος της με ίδια μέσα. Να επανέλθω σε αυτό που είπατε για τη Ρωσία. Τα, τα υποστηρίζω όλα αυτά που είπατε, συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε κοινή στάση ε, ε απέναντι στη χώρα αυτή και να συνεχίσουμε να στέλνουμε σαφή μηνύματα. Θα ήθελα όμως να μεταφέρετε στους ανωτέρους σας ε, και μια ακόμη θέση. Εμείς επιμένουμε στη συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο να τεθεί, ε, να αμφισβητηθεί η συμφωνία αυτή. Και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ο Αμερικανικός Πρόεδρος αγνοεί εννέα μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού ε, για τα Πυρηνικά που επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν τηρεί τη συμφωνία. Δεν νομίζω ότι βοηθά όταν ε, καταγγέλουμε το Ιράν για τη στάση του στην, για, στη Χεσμολά, στη Συρία, στην Ιεμένη, στους βαλιστικούς πυράβλους. Όλα αυτά είναι πραγματικά σημεία στα οποία μπορεί να ασκηθεί βάσιμη κριτική στο Ιράν. Όχι όμως η τήρηση της συμφωνίας για τα πυρηνικά. Εκεί το Ιράν έχει επιδείξει ε, εξαιρετική στάση. Ε, δεν θέλουμε στην πραγματικότητα το Ιράν να μετεξελιχθεί σε μια νέα Βόρεια Κορέα. Και δεν βοηθάει αυτή η στάση. Πιστεύω επίσης ότι και ως κράτη-μέλη αλλά και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πρέπει να ε, εντατικοποιήσουμε τις επαφές μας με τις Αμερικανικές αρχές με την Αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να κατανοήσουμε από κοινού, να, οδηγηθούμε σε μια κοινή αντίληψη για την περιπλοκότητα και τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τον, ε, τον κόσμο μας ε, και για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αξίες όπως είναι το ανοιχτό εμπόριο για παράδειγμα. Ε, έχω και ένα ερώτημα. Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή λέγοντάς του ότι έχουμε μεγάλο κατάλογο ομιλητών και ότι ε, υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικός περιορισμός. 30 δευτερόλεπτα. Ερώτημα. Έγινε η υπογραφή Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το Δεκέμβριο για την βελτίωση των ε, επιχειρήσεών μας, των αποστολών μας στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής αμήνες και ασφάλειας. Το απευθύνω στην ΕΙΕΔ. Ε, διεπηρεσιακή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες στοιχεία. ευχαριστώ. Η κυρία Λέζιν, παρακαλώ, πολύ σύντομα, για να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω και εγώ γερμανικό. Σημερίζομαι πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι προλαλήσαντες σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Έχω όμως ένα ερώτημα προς την κυρία Ράντα. Με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με συγκεκριμένες βασικές στρατηγικές των ΗΠΑ. Άκουσα στη νέα στρατηγική ασφαλείας ότι ε, διάβασα μάλλον στη στρατηγική ασφαλείας ότι η Ρωσία και η Κίνα ε, έχουν ε, μια αναθεωρητική στάση στη διεθνή σκηνή. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ε, ή επίσης συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την εκτίμηση. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εκτίμησης. Ακούγεται συχνά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία και Κίνα βρίσκονται σε ανταγωνισμό. Ναι, αλλά ανταγωνισμός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επιτιθέμεθα ο ένας τον άλλον. Άρα τι ακριβώς σηματοδοτεί και σημαίνει αυτή η ε, διατύπωση ότι πρόκειται για αναθεωρητικές δυνάμεις, για δυνάμεις που τηρούν αναθεωρητική στάση. Στην ε, στρατηγική ασφαλείας ε, το γεγονός ότι υπάρχει μια ε, εγκατάλειψη ε, της έμφασης στην αντιτρομοκρατία και μια μεγαλύτερη έμφαση σε τυχόν, σε συγκρούσεις με, με τη Ρωσία και την Κίνα. Ταυτόχρονα ανακοινώνεται η ενίσχυση του, των, των, των, των ικανοτήτων στο Αφγανιστάν. Ποιες πιστεύετε ότι, ότι θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής, κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Σου ειδικά θα μιλήσω, οπότε χρειάζεστε φαντάζομαι τα ακουστικά σας. Τρεις ερωτήσεις έχω παρακαλώ και θα είμαι σύντομη. Πρώτον, Μια ερώτηση που δεν ακούστηκε καθόλου είναι τι γίνεται τώρα ε, βόρεια της Συρίας. Η επίθεση αυτή στο Αφρίν και η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε αυτή την επίθεση ποια είναι. Οι σύμμαχοί μας ε, στο ΝΑΤΟ, έτσι. Έχει να κάνει όμως και με τη Ρωσία. Πώς ε, επεξεργάζεται το θέμα η Ρωσία. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να εγγυθείτε προσφορά ενέργειας στην Ευρώπη. Στη σελίδα 23 της στρατηγικής ασφάλειας αναφέρεστε σε ανάπτυξη ασφαλών ενεργειακών πόρων. Αν συνεχίσει όμως κανείς να διαβάζει, μετά αναφερόμαστε στα ορυκτά και όχι στις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε θέλω να ξέρω, εσείς το ξέρετε ότι εμείς στην Ευρώπη πάμε προς μια κοινωνία η οποία δεν θα χρησιμοποιεί πια ορυκτά καύσιμα. Αυτή είναι η ιδέα μας, να μην χρησιμοποιούμε πια ε, τέτοια καύσιμα στο μέλλον, αλλά μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι λοιπόν μια ερώτησή μου. Και έπειτα αναφερθήκατε στον έλεγχο των εξοπλισμών. Αλλά μόνο για τα πυρηνικά. Εμείς όμως έχουμε και άλλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και άλλα είδη ελέγχου εξαγωγών όπλων. Εμείς έχουμε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, σε διάφορους τομείς με πολύ συγκεκριμένους κανόνες για τη δυνατότητα ή όχι πώληση όπλων. Κάποιες χώρες, μάλιστα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε ακόμα πιο μακριά. Ναι, και θα ολοκληρώσω με αυτό. Θέλω να μου εξηγήσετε, να αναλύσετε κάπως την κατάσταση αυτή όσον αφορά τις χώρες τις οποίες εξάγουμε όπλα. Γιατί και εσείς όπως και εμείς εξάγουμε όπλα σε χώρες όπου τα όπλα τελικά χρησιμοποιούνται για τον πόλεμο. Σύντομοι να είσαστε παρακαλώ. Ναι, εσείς. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής, δεν τον ακούμε. Δεν ακούγεται ο μιλητής γιατί μιλάει εκτός μικροφώνου. Συγγνώμη. Λοιπόν, είδαμε τι μας είπε και ο πρέσβης σου όσον αφορά την εθνική ασφάλεια. Ότι η στρατηγική αυτή εμφανίζεται πολύ καλή στα χαρτιά, αλλά όταν δούμε τα γεγονότα της πράξης, και ο κύριος Πάιφερ έδωσε πολλά παραδείγματα, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια. Έχουμε διαφορετική εικόνα. Ένα παράδειγμα, Βόρεια Κορέα. Πριν από ένα μήνα, Ο Υπουργό Εξωτερικών είπε στο Πεκίνο, νομίζω, ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τη Βόρεια Κορέα, άπαξ και εκείνη το επιθυμεί και ευχαρίστω η πρώτη συνάντηση να γίνει χωρί όρου. μετά, μάλλον από μερικέ μέρε, ανέφερε κάποιου όρου. Από περικοποίηση, για παράδειγμα. Και ξέρουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί αν δεν έχουμε προηγουμένω συνομιλίε με την Κορέα. Και μετά εμφανίστηκε ο κύριο Τραμπ με ένα tweet που είπε ότι ο χάνει το χρόνο του προσπαθώντας να διαπραγματευτεί με μικροπατεώνες. Οπότε, τι είναι τελικά αυτή η στρατηγική. Το ένα το άλλο. Και για τη Ρωσία είπατε ότι η Ρωσία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά τους τελευταίους μήνες είδαμε ότι η Ρωσία μπλέκεται στη Μέση Ανατολή με τρόπο που για τελευταία φορά είχαμε δει τη, δεκαετία, του 60 όσον αφορά τις σχέσεις με την Αίγυπτο. Οπότε οι Ηνωμένε Πολιτείε επέτρεψαν στην Ρωσία να πάνε στη Μέση Ανατολή με αυτόν τον τρόπο που δεν είχαμε ξαναδεί τόσες δεκαετίες. Και μια ερώτηση πως την κυρία Χιντρά. Είπατε ότι οι προδιαγραφές μας της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι να αποτελεί ένα παγκόσμιο παίκτη. Θα ήθελα επιχειρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τότε τουλάχιστον που είμαι εγώ ευρωβουλευτής, λέμε ότι πρέπει να έχει μια δικιά της εξωτερική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δικιά της στρατηγική για την επίλυση κρίσεων και συγκρούσεων, ιδίω αυτών που βρίσκονται επί των πυλών μας. Με ευχαριστούμε. Λόπες Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, ξέρω μάλλον ότι γνωρίζετε τα ισπανικά. Λοιπόν, εγώ είμαι από την Ισπανία. 400 χρόνια λέγαμε πρώτα Ισπανία. Spain first. Μετά ρηπόθηκε η χώρα μας και απομονώθηκε μέχρι το 1986 που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανακαλύψαμε σε αντίθεση με κάποιους Βρετανούς, όχι όλοι βέβαια, ότι οι αυτοκρατορίες πάνε και στην Ισπανία διαπιστώσαμε ότι το να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είμαστε ένας από τους 27, μπορεί να μας βοηθήσει, ίσως όχι να είμαστε πρώτοι, αλλά αν μη τι άλλο να είμαστε ασφαλείς, προστατευμένοι. Θέλω λοιπόν να σας ε, σχολιάσω κάτι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχω να πάω κι εγώ σε άλλη συνεδρίαση, γι' αυτό και δεν κάνω ερώτηση, αλλά αυτό που θα σας ζητήσω είναι να σχολιάσετε. Ωραία, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε καλούς πρέσβεις, εσείς είσαστε ένας, αλλά μεταφέρετε αυτό στις Ηνωμένε Πολιτείες. Είχαμε δύο πρέσβεις πριν, τον και τον Κάνερ, που ήταν εξαιρετικοί Αν ήσασταν εσείς, εντάξει, τόσο το καλύτερο, αλλά χρειαζόμαστε καλούς πρέσβεις, γιατί δημιουργούνται πολλές παρεξηγήσεις με τον σημερινό πρόεδρο, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Και τα ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης, αλλά κάποιοι ρεπουμπλικάνοι στο παρελθόν είχαν κάποιου περιορισμού. Εδώ οι ευρωβουλευτέ τουλάχιστον μπορούμε και μιλάμε ελεύθερα. Λοιπόν, τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μπουστινάρου. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άνταμ και ένα πληρωτή επικεφαλή τη Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή τη συνάντηση, αυτή τη συζήτηση μετά από τα έγγραφα αυτά και θα ξεκινήσω δηλώντα το προφανές ότι η κοινή μα ασφάλεια, ΙΠΑΕ, σχετίζεται άμεσα με τόσους πολλούς τρόπους, ίσως πολύ περισσότερους από αυτούς που αποδεχόμαστε και η κοινή μας ασφάλεια έχει επιπτώσεις σε κάθε σημείο του πλανήτη. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μια κοινή ευθύνη σε σχέση με την παγκόσμια σταθερότητα να κατονομάσω μόνο κάποιους τομείς όπου η ασφάλειά μας πρέπει να είναι συνεργατική και συντονισμένη. Όπως κάναμε με την ε, διάσκεψη στο Βουκουρέστι για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια που αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για να ενισχύσουμε αυτή την δυνατότητα συντονισμού και συνεργασίας για την ε, άμυνά μας. Θα μπορούσα να φέρω και άλλα στοιχεία. Τρομοκρατία. Εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Και Δυτικά Βαλκάνια, εκεί που χρειάζεται μέγιστη συνεργασία. Συνάδελφε, τέλειωνε επιδεινώση της κατάστασης επίσης σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα πρέπει να έχουμε ενδεχομένω μονομερείς ε, δράσεις στη Μέση Ανατολή, στα πυρηνικά του Ιράν, γιατί κάνοντας το αυτό, μονομερώς αυτοί αποδυναμώνουν την παγκόσμια ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Λίτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίτς λέγουμε, από τη Γερμανία. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Όπως είπε ο κ. Γκάλερ, χαίρομαι που το ΝΑΤΟ θεωρείται μια γέφυρα και μια πηγή ασφάλειας. Σε αυτή λοιπόν την κοινή μας προσέγγιση για την άμυνα στην Ευρώπη, μήπως θα έπρεπε να ήταν καλό και γιατί είπα να έχουμε έναν αρμονισμένο σύστημα οπλικό και να δούμε ακριβώς τι γίνεται με μας εδώ. Μετά, στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, ο πρόεδρος αφαίρεσε την κλιματική αλλαγή. Εγώ μόλις πήγα στην ε, Ουάσιγκτον, μίλησα με άτομα από το Brookings, συζητήσαμε κάποια θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, κλίματος. Οπότε μήπως θα έπρεπε να μιλήσουμε και για κλιματική διπλωματία και να το θεωρήσουμε σε ένα ζήτημα το οποίο συμβάλλει στην άμυνα. Δηλαδή να αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα. Ε, πρόεδρος, ε, ε και εγώ θα πρέπει να σας ζητήσω να συντομεύετε. Ναι, θα σταματήσω εδώ και προσβλέπω στα απάντηση σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Μπούχνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κ. Μπουχνερ. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά που συμβαίνουν είναι και λίγο αντιπαραγωγικά, γιατί ενδεχομένω αποτελούν απειλή για την ειρήνη. Τι γίνεται με το Ιράν, ας πούμε, και τα θέματα ασφαλείας εκεί. Και αυτό σχετίζεται και με μια παρατηρήση του κυρίου Γκάλερ. Υπάρχει ένας τρόπος προσέγγισης των δηλώσεων του Προέδρου των είπα. Η Ευρώπη μπορεί να έχει εμπορικές σχέσεις με το Ιράν παρακάμπτοντας τα οικονομικά προβλήματα. Βεβαίως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί τα πάντα είναι να τα ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε την οπτική της στρατηγικής ασφαλής στον ΗΠΑ. Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο από ποτέ η έννοια των φιλελεύθερων δημοκρατιών, τα fake news, τι απόψε έχουμε για το Russia Today. Νομίζω λοιπόν δεν θα πρέπει να προσφέρουμε επιχειρήματα σε αυταρχικά καθεστώτα για να αποδυναμώνουν την έννοια των φιλελεύθερων δημοκρατιών και ιδιαίτερα τις κοινή μα θέση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά πόσο υπερισχύουν όσον αφορά οι εμπλέκοντες στην στρατηγική ασφαλεία των ΗΠΑ. Γιατί έχουμε ελάχιστους εταίρους που μάχονται για αυτά. Και μετά Θέλετε να μου σχολιάσετε το θέμα της συνεργασίας Ένωσης ΝΑΤΟ κατά πόσο συμβάλλει στην γενικότερη εικόνα που έχουν στην Ουάσιγκτον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στους ηγητές μας, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω και να πω ότι ως συγγήτρια του θέματος για την αντιμετώπιση της στρατηγικής, της επικοινωνικής της Ρωσίας. Να επενθυμίσω τους κύριους στόχους της επικοινωνικής στρατηγικής της Ρωσίας. Δηλαδή, η αποδυνάμωση του διατλαντικού δεσμού μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης, Καναδά κλπ. Πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού και να ενισχύσουμε τις αντίστοιχες στρατηγικές μας για αυτό το θέμα. Είχαμε μια κοινή επίσκεψη στην ΑΦΕΤ. Πήγαμε στο Norfolk, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, στη Βιρτζίνια δηλαδή και στην Ουάσιγκτον επίσης και είχαμε αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και αμερικανική αντιπροσωπεία και ακούγοντας για αυτή τη στρατηγική βλέπω ότι υπάρχει μια απόρριψη της προσέγγισης. Δηλαδή, καταρχάς, πρέπει να δούμε τι γίνεται με το άρθρο 5 και τη λειτουργία του, το άρθρο 5 της Εθνικής της Ουάσιγκτον, που μιλάει ανοιχτά για αυτά τα θέματα και προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποιες ενσυχίες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχει και το θέμα της εικόνας που έχει η Ρωσία ανάλογα με τη χώρα της Ένωσης. Αλλά τέλο πάντων όλους μας ανησυχούν οι πολιτικές, οι ρωσικές. Και εδώ η πολιτική των ΗΠΑ έχει τεράστια σημασία, είναι ξεκάθαρη, όπως και η εθνική στρατηγική. Δεν είναι θέμα εγγράφου, είμαστε αρκετά έμπειροι, αρκετοί από εμά και παρακολουθούμε καθημερινά τα αμερικανικά διπλωματικά τεκτενόμενα. Έχουμε στην σχέση με τις ΣΥΠΑ και από αυτή την άποψη είπα ηγούνται. Είναι ένας ηγέτης όσον αφορά την προστασία χωρών και κοινωνιών που κινδυνεύουν από την επιθετική πολιτική της Ρωσίας που είναι σχεδόν υπεριαλιστική. Εδώ και περίπου 10 χρόνια έτσι δεν είναι κάτι το νέο αυτό. Δεν αφορά δηλαδή την επίθεσή του στην Ουκρανία υπάρχει μια σειρά ολόκληρη γεγονότων που έχουν λάβει χώρα νωρίτερα και που έχουν κάποια συνοχή. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μια πιο συνεκτική πολιτική και εδώ και αλλού. πρέπει βεβαίως να είμαστε ρεαλιστές και να αντιμετωπίσουμε τις επιθετικές ε, τακτικές των Ρώσων σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβαμένες και της δικής μου. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε και το Ιράν. Πήγαμε στην Ουάσιγκτον. Είχαμε αυτή την διπλωματική προσέγγιση και από την πλευρά της Ένωσης και από την πλευρά των είπα για την διατήρηση του JCPOA. Αλλά δυστυχώς πρόσφατα είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και αλλού και θυμάμαι και εγώ ίδια είχα αμφιβολίες για το GCPOA στην αρχή. Αλλά μετά τη συμφωνία η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Πρέπει να δούμε πάντως το Ιράν στο σύνολό του. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι τώρα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, γιατί ήταν κοινό σημείο συζήτηση στο Ιράν μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης. Δηλαδή, σημαίνει ότι αυτό ότι είχαμε πολύ θετικές εξελίξεις μετά από τη δική μας επίσκεψη, μάλιστα. Νομίζω δηλαδή ότι η ασφάλεια η συνιστόσα της ασφάλειας και η ασφάλεια ίδια σχετίζονται με αυτή την στατηγική. Πρέπει δηλαδή να το λάβουμε υπόψη μας σε όλα αυτά που λέμε σε κάθε συνάντηση. σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Το 2003 τώρα έχουμε άλλες προκλήσεις. Και στα αριστερά του συνόρου μας και βλέπουμε και άλλα προβλήματα στα σύνορά μας κοντά. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Οπότε αυτό το νέο όραμα είναι απαραίτητο. Και όταν μιλάμε για διπλωματία του Twitter, εγώ έστω παρόδο είμαι πολύ συντηρητική και δεν το χρησιμοποιώ, γιατί νομίζω ότι είναι υπερβολικά γρήγορο εργαλείο σε σχέση με τις διπλωματικές σχέσεις. Όμως βλέπω ότι ο ίδιος Ομπάμα το είχε πρόθεση και το χρησιμοποιούν και αρκετοί ηγέτες της Ένωσης. Έτσι. Είναι πολύ γρήγορο εργαλείο. Ε, για μένα όμως το συνεχίζω, να το θεωρώ πολύ συντηρητικό. Επειδή οδηγεί σε παρανοήσεις, ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εξέχοντες ε, εισηγητές μας και Σόπφερ, ε, πρεσβευτά Σόπφερ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ πολύ τα σχόλιά σας για την στρατηγική επικοινωνία της ε, Ρωσίας. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί τη είπα και την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 70 χρόνια μας απασχολεί αυτή η στρατηγική επικοινωνία. Υπήρχε και το ράδιο ελεύθερη Ευρώπη, αντιμετωπίσαμε από κοινού το σιδρούν παραπέτασμα, έχουμε μια κοινή αντίληψη για το τι σημαίνει ελευθερία και δυστυχώς επανερχόμαστε σε μια κατάσταση που ε, επαναφέρει ορισμένα από τα ζητήματα που μας είχαν απασχολήσει βεβαίως και στο παρελθόν, χρειάζεται όμως να τα δούμε με μια νέα ματιά ε, και ε, νομίζω ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία σε αυτό το πεδίο. Θέλω να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Χαιρετίζουμε όλοι το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στο, στην, στο Bretton Woods, στην ε, συνένεση της Ουάσιγκτον. Βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια και, τα, και οι εποχές έχουν αλλάξει. Ε, ο, η Κίνα, για παράδειγμα, παίζει έναν νέο ρόλο στον κόσμο. Δεν είμαι ειδικό, αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλέ να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ε, προφανώς μια στρατηγική απάντηση ε, πρέπει να λάβει υπόψη και αυτά τα, ε, τα διαφορετικά ε, δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Και βεβαίως έχουμε μια, ένα ολόκληρο πλωστάσιο όχι μόνο τις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, ή τη στρατιωτική δύναμη, υπάρχουν, υπάρχει και η οικονομική πολιτική, υπάρχουν και οι πολιτισμικές ανταλλαγές. Φυσικά έχουμε μια μακρά παράδοση διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού συζήτησης. Αλλά ποτέ πριν από το 2014 δεν, είχε, δεν είχαν ξαναλλάξει τα σύνορα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό έγινε μόλις το 2014 ξανά. Και για, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Τώρα, αν οι απόψεις θα εκφραστούν σε επίσημα έγγραφα ή ακόμη κάποιες φορές και στο Twitter, αυτό είναι δευτερεύουσα σημασίας. Αυτό που είναι σημασία είναι ε, ότι ε, οποιαδήποτε αδυναμία ε, δική μας αξιοποιείται από τους αντιπάλους μας. Φάνηκε αυτό στην Κρυμαία το 2014 και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ε, γρήγορη, ε, γρήγορο χρόνο αντίδρασης. Ε, όπως ήταν και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία. Αν και η ενότητα που τελικά επετεύχθη μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού χρειάστηκε πολύ χρόνο για να σμιλευτεί. Βλέπω τώρα, για παράδειγμα, ότι κάθε χρόνο οι κυρώσεις επεκτείνονται και παρατείνονται με πολύ μεγαλύτερη ενότητα και με πολύ λιγότερες διαδικασίες. Και μια τέτοια στάση ε, νομίζω ότι είναι επιτεύξιμη και στο, και στο θέμα της Ρωσίας αλλά και στο Ιράν και σε άλλα θέματα. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι διατλαντικές σχέσεις δεν αφορούν μόνο κυβερνήσεις. Είναι μια πολύπλευρη σχέση που ε, περιλαμβάνει και τις ε, ε, πολύ έντονες σχέσεις που έχετε εσείς μεταξύ σας. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν περισσότερες, περισσότερα ταξίδια προς την Ουάσιγκτον ή προς τις Βρυξέλλες από κοινοβουλευτικούς και από ε, μέλη του Κογκρέσου. Ε, και βεβαίως όλα αυτά αποτελούν ομάδες εργασίας υψηλού επίπεδου. Εγώ, υπάρχει, εγώ γνωρίζω, έχω έναν κατάλογο αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν κάθε εβδομάδα στις Βρυξέλλες προκειμένου να, ε, ε, να συζητούμε θέματα ασφαλείας και άμυνας. Υπάρχουν ε, αξιωματούχοι οι οποίοι περνούν εβδομάδες ολόκληρες εδώ, Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μάλιστα επισκέπτονται και μια σειρά από πρωτεύουσες προκειμένου να συζητούμε αυτά τα θέματα. Για την Πέσκο που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο ε, Εμεί θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική απόφαση και ε, ορθή, ε, τη χαιρετίζουμε αλλά πρόκειται για μια απόφαση η οποία προς το παρόν παραμένει στα χαρτιά δεν έχει συγκεκριμένες πρακτικές επιπτώσεις ακόμα η απόφαση αυτή πρέπει να εξεταστούν θέματα διαλειτουργικότητας, κινητικότητας και για την κλιματική αλλαγή ε, να πω ότι ο κύριος Λίτς είπε άλλωστε ανέφερε αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος εξέφρασε τη γνώμη του ε, για την Συμφωνία των Παρισίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΙΠΑ δεν ανησυχούν για το περιβάλλον. Ε, μπορεί να μην είμαστε τόσο προηγμένοι όσο κάποιες χώρες της Ευρώπης για τα, όσον αφορά τα νέα καύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τα υβριδικά αυτοκίνητα. Νομίζω όμως ότι η αναφορά στα, στις καθαρότερες ε, ορυκτές μορφές ενέργειας ε, αφορά κυρίως ε, το φυσικό αέριο. Ε, εμείς τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε καταστεί σημαντικός παραγωγός φυσικού αερίου με εξαγωγές μάλιστα. Και αυτό είναι ένας, ένας παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί από τη δική μας πλευρά. Μιλώντας για την ενέργεια πάντως, οι ΙΠΑ πάντοτε υποστήριζαν την Ενεργειακή Ένωση εδώ στην Ευρώπη. Πιστεύουμε σε αυτήν, πιστεύουμε στη διαφοροποίηση του, των, των ενεργειακών πηγών. Το μείγμα βεβαίως ε, πρέπει να επιλεγεί από τις ίδιες χώρες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην εξαρτώμαστε από ένα παραγωγό και ξέρουμε όλοι σε ποιον αναφέρομαι. Κύριε Λόπες Βάιτ, ε, έχει φύγει. Ε, δεν είμαι πρέσβης, αλλά μπορώ να σας απαντήσω στα ερωτήματα που θέσατε και κατα, κατηδίαν μπορούμε να ε, οργανώσουμε συναντήσεις, αν κάποιος ενδιαφέρεται από εσάς, προκειμένου να μπορέσουμε να φωτίσουμε περισσότερα, περισσότερα τα ζητήματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν ε, και να μιλήσουμε και για την άξα, για τη συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν με ρωτούσατε πριν από 5-10 χρόνια, ε, αν πίστευα ότι θα υπήρχε η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ που ξέρουμε σήμερα, θα απαντούσα όχι. Δεν είναι κάτι που το περίμενα. Φυσικά ε, είναι απολύτως λογική αυτή η συνεργασία. Έχουμε την, ε, την έδρα μας και οι δύο οργανισμοί ε, στην, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει ένας, μια ολόκληρη γκάμα ε, θεμάτων στα οποία συνεργάζονται τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ αλλά υπάρχουν και πολλά, πολλά, πολλά νέα θέματα όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, η Ρωσία, η Κίνα, η Ανατολική Εταιρική Σχέση, οι απειλές ε, που ε, έχουν αναδειχθεί σε μια σειρά αποτομής αλλά και μια αντίληψη ότι μέσα από την κοινή ανάληψη ευθυνών μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα κοινά μα συμφέροντα. Είναι πραγματικά εκπληκτική η πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το θέμα. Να δω λιγάκι τι σημειώσει μου. Για την JCPOA και, την και για την Βόρεια Κορέα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, όμως Πρόκειται για θέματα τα οποία τα επεξεργαζόμαστε ακόμα. Ξέρετε ποια είναι η στάση μας. Μας ανησυχεί πάρα πολύ ο ρόλος του Ιράν. Αν μάλιστα δείτε τις πρόσφατες συνομιλίες που είχαμε με, τη, με τους συναδέλφους ε, στο Άρι 3 και, με την, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι φωτίζεται καλύτερα πόσο περίπλοκα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ε, σε αυτό το τμήμα του κόσμου. Για τη Βόρεια Κορέα και αυτό το θέμα ε, χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις. Υπάρχει διάλογος, υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ ΙΠΑς, ε, ΙΠΑ και ναι, Βόρειας Κορέας. Ξέρω ότι υπάρχουν αντίστοιχοι διάβλοι επικοινωνίας και μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Τον πυρηνικό αφοπλισμό της ε, Βόρειας Κορέας. Ελπίζω να τον κατακτήσουμε αυτό το στόχο. Η στάση της Κίνας ε, ήταν επικοδημοτική και χρήσιμη. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, βεβαίως. oh, yes. Για το κλίμα. Ε, ξέρετε, η ιστορία αυτή με το κλίμα... Εμείς εξακολουθούμε συμμετέχουμε σε ε, επιτροπές που συστάθηκαν με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων εμείς αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μας. Και παραθέτω τον Μάικλ Μπλουμπέργκ που είναι θερμός υποστηρικτής ε, των συμφωνιών του Παρισιού. Η αποχώρηση της κυβέρνησης δεν σημαίνει ότι ε, δεν, μπορούμε να να συνεχίσουμε τη συνεργασία ή δεν μπορούμε να θέσουμε και δικούς μας ε, στόχους που προσυδειάζουν σε εκείνους των, των Παρισίων. Ναι, είμαστε όμως ε, μια μεγάλη χώρα, διαφορετική χώρα, ε, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ε, και υπάρχουν παράγοντες στους οποίους εμείς πρέπει να συνυπολογίσουμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάνει ενδεχομένως η, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και ε, παραγωγή λιγνίτη σε ορισμένες πολιτείες μας. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να εγκαταλείψουμε εμείς με τον ίδιο ρυθμό τουλάχιστον που το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που περνάει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, υδροηλεκτρισμό κτλ. κτλ. Είναι γεγονός ότι και εμείς προς την ίδια κατεύθυνση κινούμαστε, ε, θέλουμε και με, να ε, προσφέρουμε εναλλακτικές πιο καθαρές ως προς την ενέργεια στους καταναλωτές μας, βεβαίως. Πρόεδρο, συγγνώμη που πρέπει να παρέμβω, αλλά βλέπετε έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Παρακαλώ κυρία Γκρά. Ωραία, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και επειδή ακούσαμε ότι θέλουμε και εμείς να είμαστε συμβατοί με την ε, αντιπροσωπεία των ΗΠΑ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνοπτικά στις ερωτήσεις σας. Όλες αυτές οι αλλαγές την κυβέρνηση, λέμε ότι πρέπει να δούμε τι λένε, τι από αυτά που λένε γίνονται και αντίστοιχα και εμείς να δούμε πώς θα πρέπει όχι να προσαρμόσουμε τις δικές μας πολιτικές. Πρέπει να πω ότι πραγματικά συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένε Πολιτείες πάρα πολύ καλά και ξέρουμε πόσο ζωτική σημασία είναι αυτή η σχέση, είτε για την ασφάλεια, είτε για την άμυνα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει επίσης να πω ότι στα θέματα ασφάλειας η συνεργασία τώρα είναι πιο έντονη από ό,τι κατά το παρελθόν και το είπε και ο Άνταμ. Τόσες επισκέψεις, τόσες ανταλλαγές, τόσες δεσμεύσεις του ενός προς τον άλλον να κατέρθουν τον Ατλαντικού είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο σχέσεις με την Ουάσιγκτον, είναι σχέσεις και με διάφορα think tanks απανταχού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ερευνητέ, με εμπόριο, business. Βλέπουμε λοιπόν, το αποδεικνύεται αυτό και από τις περισσότερες εμπορικές συναλλαγές που έχουμε μεταξύ μας. Τώρα συμφωνούμε με την πολιτική. Πάντως υπάρχουν θέματα με την Κίνα εμπορικά και χάρη σε πολλούς συναδέρφους τα αντιμετωπίσαμε. Ρωσία, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Αυτά είναι θέματα με τα οποία δεν συμφωνούμε ή που η δικιά μας πολιτική τέλο πάντων είναι διαφορετική από εκείνη των ΗΠΑ. Το JCPOA και άλλα. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάθε φορά συντονισμό και να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει στις αρχές και τις αξίες της και στη δικιά της πολιτική και να πούμε ότι, συγγνώμη, μπορεί η Αμερικανική πολιτική να είναι κάπως διαφορετική από τη δικιά μας, αλλά η δικιά μας αυτή είναι. Και ας κοιτάξουν αλλού για συμμάχους. Να επαναλάβω επίσης το ότι προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους και ο κύριος Λίτς αναφέρθηκε σε αυτό. Συνδυασμό ασφάλειας και κλίματος. Φυσικά και υπάρχει ευρύ πεδίο για συνεργασία που σιγά σιγά ανακαλύπτουμε και εμείς νέους τρόπους και αυτό σημαίνει νέος τρόπος σκέψης, νέα προσέγγιση στις σχέσεις μας και νέα θετικά ζητήματα στη σχέση αυτή εξαιρετική συνεργασία έχουμε στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, πολύ περισσότερο τώρα από παλιότερα, ενέργεια, ενεργειακά ζητήματα. Και εδώ άλλο ένας τομέας στον οποίο θέλουμε ακόμα περισσότερη συνεργασία. Οπότε είναι θετικά όλα αυτά. Πρέπει να δούμε βέβαια την εθνική στρατηγική και να αντιδράσουμε σε αυτή. Πρέπει να δούμε την ε, στρατηγική άμυνας και να αντιδράσουμε. Αυτό είναι ο δρόμος, αυτό κάνουμε και είναι πολύ καλό που βρισκόμαστε και ακόμη και τις δικές σας ε, απόψεις, γιατί οι κοινοβουλευτικές σχέσεις με το Κογκρέσο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κυρίως τη σήμερον ημέρα, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σχέση μεταξύ μας. Ευχαριστούμε, ο πρέσβης Πάιφερ. Ευχαριστώ πολύ να σχολιάσω και εγώ διάφορα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, να σχολιάσω για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλεια. Είναι ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο και σε αντίθεση με πολλά κυβερνητικά έγγραφα που λένε κάντε τα πάντα, αυτή η στρατηγική θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Χάρη στον Υπουργό. Τώρα, ε, λόγια και πράξεις. Όντως, αυτά που ακούσαμε από τη Ουάσιγκτον μερικέ φορέ ήταν, προκαλούσαν σύγχυση, αλλά δούμε τις πράξεις, τα έργα. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, αυτά που είπε ο πρόεδρος, αλλά οι Αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να συνεργάζονται με την Ευρώπη όπως το ξέρουμε και έχουμε συμφωνήσει ήδη από το 2016 παρόλο τα όσα έχει πει ο πρόεδρος στην προεκλογική εκστρατεία του και μετά βλέπετε επίσης μεγάλη συνεργασία για θεματα ρωσια Ρωσία-ουκρανία. Όσον αφορά τα tweets είναι ένα πράγμα που ζητήσαμε να αλλάξει δεν θα γίνει όμως. Τι να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε με ό,τι έχουμε. Μέχρι τώρα είχαμε επιτυχία στην πολιτική μη διάδοσης των πυρηνικών. Αυτό πάντως που ο πρόεδρος κάνει είναι ότι έχει τα δικά του ζητήματα. Τώρα, με ρωτήσατε υπάρχουν άλλοι τρόποι χωρίς να αλλάξουμε τη συμφωνία JCPOA. προσπαθούμε τις δεσμεύσεις να τις σφίξουμε κάπως. Αυτό. Για τη Βόρεια Κορέα είναι τυχές που ακούμε διαφορετικά λόγια από τον Υπουργό και διαφορετικά από τον Υπουργό για το πώς να διαπραγματευτούμε με τη Βόρεια Κορέα. Αυτό αντικατοπτρίζει σε ένα βαθμό το γεγονό ότι ο Άσιγκτον προσπαθεί να έχει μια σκληρή προσέγγιση απέναντι στη Βόρεια Κορέα. Και μετά έρχεται το ερώτημα, η ίδια η Βόρεια Κορέα τι θέλει. Άλλοι λένε ότι θέλουν τα πυρηνικά για να αποτρέψουν επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι και η κυβέρνηση των Ηνωμένων λέει όχι, θέλει τα πυρηνικά για κάτι παραπάνω για να βγάλει από την Κορεατική Χερσόνησο τις Ηνωμένες Πολιτείες πλήρως. Και αν το δείτε έτσι βέβαια είναι αλλιώ. Οπότε αυτά που ακούγονται είναι διαφορετικά. Γιατί, Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει η Βόρεια Κορέα. Και τέλος για το κλίμα. Ήταν σφάλμα για τις ΗΠΑ να αποσυρθούν από την κλιματική συμφωνία. Όμως, δείτε τι κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των διαφόρων πολιτιών. Κάνουν πράγματα. τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και όσον αφορά για το κλίμα και την ασφάλεια, το σχόλιο μου είναι ότι λίγοι φορείς σκέφτονται ότι μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα στρατιωτικά. Ό,τι διαφωνίες προκύψουν θα πρέπει βέβαια στο μέλλον να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές μας για αυτήν ε, τη συζήτηση που είχαμε όσον αφορά την εθνική στρατηγική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, οπότε να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε. Παραμείνετε, διότι έχουμε την επόμενη πολύ σημαντική συζήτηση που θα ακολουθήσει και που είναι η συνθήκη INF για τα πυρηνικά όπλα μέσου Ελληνικούς. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, οπότε θα αρχίσουμε. Ξέρω ότι πήρε πολύ χρόνο η προηγούμενη συζήτηση, ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά έχουμε εξίσου σημαντικό θέμα τώρα να εξετάσουμε. Πρόκειται για τις ε, δυσκολίες στην εφαρμογή της συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσω Και είναι προνόμιο για μένα και ιδιαίτερη χαρά να υποδεχτώ εδώ τους ομιλητές μας. Πρώτα απ' όλα τον Σεντ Μπιλίτσα που σας είναι γνωστός. Έχει έρθει και ξανάρθει εδώ είναι ο ειδικό απεσταλμένο για τον αφοπλισμό και την μη διάδοση. Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση και τμήματάρχη στη ΣΕΚΠΟΛ 1. Δεύτερος ο μα θα είναι ο κύριος Βίλιαμ Αλπέρκε, ο οποίος είναι στο ΝΑΤΟ, στο κέντρο του ΝΑΤΟ, που ασχολείται με τον αφοπλισμό και την μη διάδοση. Ίσως δεν τα λέω με τη σειρά όσον αφορά το όπλο μαζικής καταστροφής και τον έλεγχο των εξοπλισμών. Ίσως δεν τα με τη σωστή σειρά τις ιδιότητές σας, αλλά πάση περιπτώσει ελπίζω να σας περιέγραψα σωστά. Όσον αφορά τα καθήκοντά σας και τις αρμοδιότητές σας. Και ο τρίτος, ο πρέσβης Στίβεν Πάιφερ και πάλι, ο οποίος είναι ανώτερος εξωτερικός ε, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Brookings στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η συνθήκη αυτή μας απασχολεί για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνικούς και οι δυσκολίες της. Πρώτα απ' όλα το λόγο στον πρέσβη Μπλίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την Επιτροπή σας για την θαυμάσια προηγούμενη συζήτηση για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλεια στον ΗΠΑ, που ήταν πολύ ενημερωτική για πολλούς από εμά που την ακούσαμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για αυτή τη συνάντηση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και είναι τιμή μου που συμμερίζομαι την παρουσίαση με θαυμάσιους συναδέλφους εδώ από τις Βρυξέλλες και το Ινστιτούτο Μπρούκινγκ στη Ουάσιγκτον. Καταρχά στα πρώτα μου σχόλια να αναφερθώ σε τρία κυρία σημεία. Καταρχάς, βασικές πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουμε, κάποιες αλλαγές και προκλήσεις για αυτή τη συνθήκη μετά από 30 χρόνια ύπαρξης και η θέση της ΕΕ σε σχέση με αυτή την συνθήκη και άλλα σχετικά ζητήματα. Καταρχάς τα βασικά στοιχεία για την ε, συνθήκη μεταξύ ΙΠΑ και ΕΣΟΣΟΔΟΥ για τον περιορισμό μέσου και μικρού βελληνακού. Καταρχά είχε υπογραφεί από τον Κορπατσόφ και το Ρίγκαν το 1987 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1988. Και οι δύο χώρε είχαν την υποχρέωση να εξαλείψουν όλους τους βαλιστικούς ε, πυράβλους και τους πυράβλους κρούς από τα 500 μέχρι τα 5.500 χιλιόμετρα. Για πρώτη φορά οι υπερδυνάμεις είχαν συμφωνήσει δηλαδή να μειώσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο εξαρτώντας τελείω μια ολόκληρη κατηγορία πυρηνικών όπλων. Μετά από εντελεχείς ελέγχους και επισκέψεις στις τοποθεσίες εκτόξευσης. 2.600 ε, ε, κεφαλές είχαμε που εξαφανίστηκαν μετά την ε, εφαρμογή της συνθήκης μέχρι τον Ιούνιο του 1991. Μετά από τη διάλυση της ΕΣΕΣΟΔΟΥ του 1991, η Ρωσική Ομοσπονδία αποτέλεσε τον διάδοχο εταίρο σε αυτή τη συμφωνία και τον Οκτώβριο του 2007 πρότεινε η Ρωσία μια, μια πρωτοβουλία για να προσθέσουμε μια συνολικότερη διάσταση σε αυτή τη ε, συνθήκη πρότεινε ότι αυτή η διμερή συμφωνία να μετατραπεί σε πολυμερή συμφωνία και η διάσκεψη στη Γενέβη το 2008 είδε να παρουσιάζεται από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών μια νέα, ένα νέο πλαίσιο συμφωνία για την ε, μείωση του μέσου και ε, μικρού ελληνικού πενικά όπλα. Που ε, σύμβαση η οποία ήταν ανοιχτή και, και σε άλλου. Για πρώτη φορά υπήρχε στήριξη αυτή την ιδέα. Υπήρχαν βέβαια και άλλε προτάσει για τέτοιου είδου συμφωνίε και σε άλλε περιοχέ του κόσμου που βασίζονταν στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Σε αυτό λοιπόν το υπόβαθρο οι προπαρασκευαστικές επιτροπές του 2008 αξέδωσαν μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται τα εξής. Καλωσορίζουμε την συνεχή υποστήριξη για αυτή τη συμφωνία στην 62η διάσκεψη του ΟΗΕ και καταγράφουμε την συζήτηση και την πρόθεση για τον περιορισμό όλων των μικρού και μεσαιοβελληνικών πυρηνικών όπλων. Σε αυτό το πλαίσιο είχε καταγραφεί επίση και η πρόταση η γαλλική του Μάρτιου 2008 για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει για την απαγόρευση των πυραυλών εδάφους μικρού και μεσαίου βελνικού. που όμως τελικά δεν εφαρμόστηκε. Το Ιούλιο του 2014 η ΕΠΑ ε, κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι παραβίασε αυτή την ε, συνθήκη επειδή ακριβώς δεν έδωσε στοιχεία όσον αφορά τα σημεία εκτόξευσης πυράβλων εδάφους εδάφους μεσαίου ή μικρού βελληνικούς και η αξιολόγηση που ακολούθησε από το Υπουργείο Εξωτερικών το 2016-2017 τον είπα συνέχισε να αναφέρει αυτές τις, ε, αυτούς τους ισχυρισμού, ότι δηλαδή η Ρωσία συνέχισε να πειραματίζεται με αυτού του είδους όπλα και υπήρξαν εκθέσεις ότι πραγματικά η Ρωσία είχε τοποθετήσει τέτοιου είδους ε, πυρηνικά όπλα. Η Ρωσία βεβαίως αρνήθηκε ότι παραβίασε αυτή τη συμφωνία και ε, ισχυρίστηκε ότι οι είχαν κάνει το ίδιο, ότι είχαν κάνει αυτή την παραβίωση με τοποθέτηση όπλων στην ε, Ρουμανία και στην Πολωνία. Είχαμε μια ειδική επιτροπή επαλήθευσή, όπως ακριβώς προβλέπει το άρθρο 13 της Επιτροπής, που προβλέπε και δημιουργήσει επαφέ μεταξύ ΙΠΑ και Μόσχας. Στην Γενέβη, το Δεκέμβρη πέρσι είχαμε μια συνάντηση όπου αντιπροσωπείε από Καζακστάν, Λευκορωσία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ουκρανία συναντήθηκαν για να συζητούν θέματα τα οποία αφορούν την εφαρμογή των υποχρεώσεων Τη ε, συνθήκη αυτή και εξέδωσαν μετά μια δήλωση προ τα ΜΜΕ κατά στο εξή. Μετά από την 30η επέτειο της υπογραφή τη συνθήκης για την προσωπία, εξέφρασε την άποψη ότι αυτή η συνθήκη θα να διανοματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με την διεθνή ασφάλεια, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση. Να τονίσω όμως ότι το άρθρο 12 της συνθήκης αυτής αναφέρει ότι τα συμβαλόμενα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικά μέρη για να επαληθεύσουν την ε, τήρηση των αμφωτέρων μερών ή όλων των μερών της συνθήκης αυτής. Στις 8 του Δεκέμβρη πέρσι η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των ρωσικών παραβιάσεων και ε, αυτό θα είναι βεβαίω και το αντικείμενο των ε, εισηγήσεων των συναδέλφων εδώ στο πάνελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτή η συνθήκη δεν ε, αποτελεί μόνο, όπως αναφέρει το πρωί, μια συμβολή στην παγκόσμια ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα και στην τήρηση του άρθρου 6 αλλά συμβάλλει και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την ασφάλιση του ότι θα παραμείνει η Ευρώπη ελεύθερη ήπειρος από οποιαδήποτε παρουσία πυρηνικών όπλων, τα οποία ήταν μέχρι τώρα ήταν ε, χιλιάδες και οι οποίες, τα οποία ήταν χιλιάδες και τα οποία όμως παραμένουν σε χώρες μέλη τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα, θα συνεχιστεί η επιτήρηση και για την τήρηση της ε, συμφωνίας και η συζήτηση αυτή τη συνθήκη σε διάφορα εθνή φόρα, στην Γενέβη, στην Επιτροπή Αφοπλισμού, σε διάφορες διασκέψεις και σε άλλες περιστάσεις. Επίσης συζητήθηκαν και οι λεπτομέρειες των διμερών διαλόγων για την μη διάδοση και για τον αφοπλισμό, εκεί όπου είχα την ε, τιμή να συμμετάσχω στις ε, επαφές αυτές μεταξύ ΙΠΑ και Ρωσία, η πιο πρόσφατη εδώ το Δεκέμβρη στις Βρυξέλλες και να σας διασφαλίσω ότι επανειλημμένω έθεσα το θέμα αυτής της συνθήκης. Και πριν από δύο μέρες, στην αρχική δήλωση για την διάσκεψη για τον αφοπλισμό στη Γενέβη, τονίστηκε το ότι η σημασία διατήρησης και συντήρησης της συνθήκης αυτής είναι είναι μεγάλη, είναι τεράστια και γίνεται έκκληση σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους γιατί αποτελεί ένα ορόσημο όσον αφορά τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων και αποβλέπει στην, στην εξά, εξάλληψη ολόκληρης κατηγορίας πυρηνικών όπλων τα οποία απαριθμούνται γύρω στις 3.000 και τα οποία είναι διάσπαρτα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αποτελεί επίσης ε, Μάλλον ε, γίνεται έκκληση επίση σε όλα τα συμβαλώμενα μέρη να τηρήσουν τι υποχρεώσει του σε δυνάμει του άρθρου 6 τη συνθήκη αυτή. Καταγράψαμε επίσης ότι μέχρι τις 5 του Φλεβάρι του 2018 η ΕΠΑ και προβλέπεται να θέσουν όρια για τα στρατηγικά όπλα για τη νέα συνθήκη START και ταυτόχρονα ενθαρρύνονται τα μέρη να επεκτείνουν τη συνθήκη και σε άλλα τμήματα του οπλοστασίου τους και στρατηγικού και μη στρατηγικού. Ιδιαίτερα ενθαρρύνουμε τις τη Ρωσία να περιλάβουν τα μη στρατηγικά όπλα στις προσπάθειες ε, ελέγχου και μη διάσωσης, όπως επίσης και να συνεχίσουν περαιτέρω συζητήσεις, ε, ελέγχους και να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο των οπλικών ε, πυρηνικών του συστημάτων για και να τα περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατόν. Ακριβώς για να περιορίσουμε και τους κινδύνους ατυχήματος πυρηνικού πολέμου υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όλα τα μέρη θα πρέπει να τηρήσουν τι υποχρεώσει όπω αυτέ προβλέπονται από αυτή τη συνθήκη για τον περιορισμό των στρατικών πυρηνικών όπλων και ε, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επίτευξη πλήρου προόδου σύμφωνα με το άρθρο 6 τη συνθήκη αυτή. Αυτή λαμβάνοντα υπόψη ότι υπάρχει ιδιαίτερη ευθύνη εκ μέρου των χωρών, οι οποίε διαθέτουν βεβαίω τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια. Εμεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ε, ομόφωνη για τον περισμό και εξάλληψη αυτού του είδους πυρηνικών όπλων. Και είναι προφανές ότι και το γράμμα αλλά και το πνεύμα αυτής της συμφωνίας είναι ύψης της ε, σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνάδελφοί μας από την Πολωνία και τις ε, κατοχώρες έκαναν αυτές τις πρώτες αξιολογήσεις. Τέλος για τους βαλιστικούς πυράβλους γενικότερα τα τεστ ανάπτυξη και χρήση βασιστικών πυράβλων από συγκεκριμένε χώρε αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίηση, δημιουργεί ε, ατμόσφαιρα δυσπιστία και αβεβαιότητα στι διεθνεί σχέσει και η επιτάχυνση ε, πυραυλικών συστημάτων στην Ασία και στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική λόγω ακριβώ των βασιστικών προγραμμάτων στην Βόρεια Κορέα, στο Ιράν, στη Συρία η ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων, στην ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους κυριότερους πρεσβευτές του κώδικα διοντολογίας για τη μη διάδοση αυτών των όπλων. Δεν απαγορεύουμε την ακριβώς διάδοση των όπλων αυτών, αλλά την περιορίζουμε ακριβώς υπέρ των χωρών που συμμετέχουν στις ηθίκες αυτές και ε, εδώ συμπεριλαμβάνεται και οι προανακοινω... Ε, προανακοινωθήσεις επεκτάς αυτών των όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μακρά ιστορία στήριξης αυτή τη συνθήκη αυτών των προσπαθειών και διπλωματικά αλλά και οικονομικά και μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβρη είχαμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπέρ αυτής της συνθήκη είχαμε την ε, γραμματεία η οποία υποστηρίζεται από την έρευνα για τι στρατηγικές έρευνε. Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερα προηγουμένως, ίσω θα ήταν ενδιαφέρον για όλα. Συγγνώμη. Η Πολωνία που έχει την ε, προεδρία της γραμματείας να πούμε ότι έχει εφαρμόσει ένα κώδικα διοντολογίας ο οποίος προωθεί την διαφάνεια και τον έλεγχο και η Πολωνία βεβαίως είναι υπέρ της πλήρης εφαρμογής αυτού του κώδικα διοντολογίας προς ενισχύση βεβαίω και των δεσμών μας με τον ΟΗΕ όπως ακριβώς τονίζει και η δήλωση και το ψήφισμα του ΟΗΕ για τα θέματα αυτά. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτά που κάνει η ΕΣΚΟΚ δεν υποκαθιστούν αυτά που γίνονται σε ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο για τον περιορισμό και την μη διάδοση αυτών των απλών. Αυτά είχα να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας για πιθανές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Σημειώσαμε όλα αυτά που είπατε, κύριε Μπιλίτσα. Και χαίρομαι που έχουμε τόσες πολλές ε, πολωνικές πρωτοβουλίες ε, στον τομέα αυτό. Κύριε Βίλιαμ Αλμπέρκ από το ΝΑΤΟ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή σας για την πρόσκληση που μου απίφθηνε. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ στο ίδιο πάνελ με τους φίλους μου, τον Γιάτσεκ και τον Στίβεν, που και οι δύο για μένα ε, είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμβαδίσει και το έργο των οποίων έχω ε, παρακολουθήσει στενά. Οι παρατηρήσεις μου ε, βεβαίως θα αφορούν την οπτική του ΝΑΤΟ για την συγκεκριμένη συνθήκη. Να ξεκινήσω ποια είναι, με το ποια είναι η απάντηση του ΝΑΤΟ ε, στην, ε, στην κρίση σε σχέση με αυτή τη συνθήκη. Τον Ιανουάριο του 2014 οι ΗΠΑ εξέφρασαν για πρώτη φορά τις ανησυχίες τους σχετικά με την παραβίαση της συνθήκης αυτής από την Ρωσία. Ε, θα είδατε ότι τον Ιούλιο του ίδιας χρονιάς ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ε, καλώντας ε, την Ρωσία να επανέλθει σε καθεστώς πλήρους συμμόρφωσης. Ε, αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2014, στη Σύνοδο του, του ΝΑΤΟ και στην σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη, καλείται η Ρωσία να ε, μην παραβιάζει και να τηρεί τη συνθήκη. το ίδιο επαναλήφθηκε σε ανακοίνωση του 2016 σε σχετική ανακοίνωση του ΝΑΤΟ. Η επιτυχία ή αποτυχία των προσπαθειών αυτών θα επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και είναι ύψης της σημασίας ε, να τηρούνται ορισμένες διατάξεις ε, που περιλαμβάνονται στη συνθήκη αφορούν τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση. Όσον αφορά τη, βιώσιμα, τη βιωσιμότητα ε, της συνθήκης, ε, αναφέρεται και η ανάγκη πλήρους επαλήθευσης της συμμόρφωσης. Ε, το Δεκέμβρη, μάλιστα, ε, υπήρξε και μια σχετική συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Γενέβη, όπου εκδόθηκε και ανακίνηση ανακοίνωση όπου τονίζονται για άλλη μια φορά οι η κρισιμότητα και η σημασία που έχει η τήρηση των συνθήκων για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών. Υπάρχει κίνδυνος η παραβίαση αυτής της συνθήκης να, να απειλήσει ε, πραγματικά την ειρήνη και την ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, υπάρχουν επίσης και νέοι πύραυλοι που αναπτύσσει η Ρωσία που ε, ε θέτουν ε, ε, που θέτουν σε κίνδυνο την, ε, την ασφάλεια στον κόσμο. ταυτόχρονα αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές ότι οι ΙΠΑ ακολουθούν και σέβονται τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους πλήρως. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί με πολλές, σε πολλές συναντήσεις και πολλές ανακοινώσεις. ο, ο έλεγχος των οπλοστασίων είναι ύψης σημασίας για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν ότι από τις ανακοινώσεις του ίδιου του ΝΑΤΟ ε, το ΝΑΤΟ παραμένει δεσμευμένο στον, στον αφοπλισμό και τη μη διάδοση και γι' αυτό το λόγο καλεί το ΝΑΤΟ τη Ρωσία να επανέλθει σε καθεστώς πλήρους συμμόρφωσης. Η ανακοίνωση του Δεκεμβρίου ε, είναι και μια υπενθύμηση προς τη Ρωσία ότι η συνθήκη αυτή δεν θα καταργηθεί και ότι η Ρωσία είναι υποχρεωμένη να έρθει σε διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και, και ιδίως της ΕΠΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εφαρμογής της. Έχει μια μακρά ιστορία. Άλλωστε, η στάση των ε, νατοικών συμμάχων στον τομέα αυτό που ξεκίνησε από το 1977 και πάντοτε βεβαίως ε, αποτελεί σημαντικό στοιχείο ο βαθμός συνεργασίας ε, με την Ρωσία ε, όσον αφορά τα θέματα της μη διάδοσης και του αφοπλισμού. Το ΝΑΤΟ επίσης έχει μειώσει δραματικά το πυρηνικό του οπλοστάσιο στην Ευρώπη. Και παρόλο που εμείς θα θέλαμε τον εφοπλισμό, είναι ακριβώς ζητήματα όπως η παραβίαση των συνθήκων από τη Ρωσία που εμποδίζουν ε, την, τον πλήρη αφοπλισμό. Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που είναι απαραίτητες ε, προκειμένου να καταλήξουμε στο στόχο του αφοπλισμού. Γιατί, θεωρώ, γιατί θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η συνθήκη. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 ε, οι αντιπαραθέσεις Σοβιετικής Ένωσης ΗΠΑ είχαν δύο στοιχεία. Πρώτον, τεράστια τεράστιες, τεράστιες στρατιωτικές μονάδες ε, εξοπλισμένες με πυρηνικές κεφαλές οι οποίες βρίσκονταν αντιμέτωπες στα σύνορα κατά μήκος του σιδηρού παραπεράσματος που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ε, τεράστια καταστροφή στον κόσμο. Ωστόσο, ε, τα, οι πύραυλοι ε, μέσου που βρίσκονταν εδώ στην Ευρώπη δεν θεωρούνταν ε, αποτρεπτικά στοιχεία ούτε θεωρούνταν εργαλεία για την εξασφάλιση της ειρήνης. Υπήρχαν μεγάλες τεχνικές δυσκολίες και περιορισμοί όσον αφορά τον ανεφοδιασμό και την, την πραγματική χρήση και ε, αξιοποίηση αυτών των ε, οπλικών συστημάτων. Ε, δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόπιστα ούτε ιδιαίτερα, ούτε ιδιαίτερα ακριβή τα οπλικά αυτά συστήματα των βαλιστικών και πυράβλων κρούζ. Οι Σοβιετικοί είχαν αντίστοιχα συστήματα εγκατεστημένα κατά μήκο των χωρών του σιδηρού παραπετάσματος οι είχαν πυρηνικές κεφάλες στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά υπήρχε ε, το, το πρόβλημα ότι ε, η ύπαρξη αυτών των πυράβλων αποτελούσε μια συνεχή, ένα συνεχή κίνδυνο ε, για την ασφάλεια και την ειρήνη. Τα οπλικά αυτά συστήματα δεν χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη ακρίβεια. Ταυτόχρονα οι ΙΠΑ είχαν υπεροπλία όσον αφορά τα ICBM, ε, και γι' αυτό δεν χρεώ... θεωρούσαν ότι δεν χρειάζονταν ε, όπλα μέσου Ε, Στη συνέχεια, στα μέσα της ε, δεκαετίας του 70, η Σοβιετική Ένωση εισήγαγε τους SS-20, που ήταν πύραυλοι μέσου βελληνικούς και τους οποίους εγκατέστησε στην Ευρώπη. Είχαν ήταν πολύ πιο προηγμένη αυτή η πύραυλη με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Και αυτό έδωσε στους Σοβιετικούς ε, τη δυνατότητα ε, να πραγματοποιήσουν προληπτικό χτύπημα χωρίς πρώτερη κοινοποίηση ε, ή προειδοποίηση του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν η, η SS-20 διάβρωσαν την αντίληψη που υπήρχε και την πεποίθηση που υπήρχε ότι ε, υπήρχε μια πυρηνική ασπίδα στην Ευρώπη του ΝΑΤΟ που προστάτευε τις ε, χώρες της ε, Ευρώπης από πιθανό σοβιετικό χτύπημα. Το 19... 80 ε, ε, πλέον ε, η πυρηνική ασπίδα του ΝΑΤΟ ήταν σχεδόν άχρηστη λόγω το, το, της στρατηγικής υπεροπλίας της Σοβιετικής Ένωσης στους βαλιστικούς πυράβλους λόγω των, των τεχνικών, της τεχνικής πρόοδου που είχαν πραγματοποιήσει εκεί. Αυτό δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και αναγκάστηκαν το ΝΑΤΟ και η ΙΠΑ και το ΝΑΤΟ να θέσουν σε καθεστώς πλήρους ετοιμότητας όλο τους το πλωστάσιο στην Ευρώπη. Και αυτό σήμαινε ότι σε μια οποιαδήποτε κρίση θα μπορούσε ε, η ένοπλη σύγκρουση να κλιμακωθεί πάρα πολύ γρήγορα σε πυρηνική σύγκρουση χωρίς να υπάρχουν ε, τα απαραίτητα ή συνηθισμένα σημάδια προειδοποίησης πριν από μια σύγκρουση. Έτσι λοιπόν ε, επρόκειτο για μια προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης να αποσυνδέσει και να διαβρώσει την ε, συμμαχία μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και ε, ΗΠΑ. Υπόθηκε ε, λοιπόν στους, ε, Αμερικανούς από τους Σοβιετικούς ότι σε περίπτωση που υπάρξει ένοπλη σύγκρουση, σύγκρουση εμείς πλέον έχουμε τη δυνατότητα να χτυπήσουμε την επικράτεια των ΗΠΑ. Η απάντηση του ΝΑΤΟ τότε ήταν ότι δημιουργήθηκε μια ε, νέα ομάδα για τον πυρηνικό σχεδιασμό. Και πρώτο καθήκον αυτής της ομάδας ήταν να προσδιορίσει τι θα γίνει και τι θα κάνει σε περίπτωση χτυπήματος από αυτούς τους ε, πυράβλους μέσου βελληνικού της Σοβιετικής Ένωσης. Κατέληξε ε, σε κάποιες συστάσεις το 1979 πρώτο βήμα ήταν να ε, εγκατασταθεί ένα σύστημα βαλιστικών πυράβλων στην Ευρώπη από το ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, ε, δεύτερη προσέγγιση ήταν να ακολουθεί μια στρατηγική για τον αφοπλισμό. Οι υπουργοί των χωρών του ΝΑΤΟ υποστήριξαν αυτές τις συστάσεις και δημιούργησαν μια ε, ομάδα ε, προκειμένου να προχωρήσουν και να προωθήσουν αυτές τις ε, συζητήσεις μέσω και δημερών σχέσεων, συζητήσεων με την Ρωσία. Και αυτό ήταν το πρόπλασμα αυτού που τελικά αποτέλεσε τη συνθήκη INF. Η συνθήκη αυτή ήταν τόσο σημαντική για το ΝΑΤΟ που οι σύμμαχοι έπρεπε να υπογράψουν αυτήν την υπογράφη αυτή την συνθήκη. Και βεβαίω ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα που θα ρωτούσαν οι Σοβιετικοί θα ήταν το ΝΑΤΟ έχει εγκρίνει αυτή την συνθήκη. Αν λοιπόν δεν είχαμε τότε δεχτεί ε, μέσω του ΝΑΤΟ να υπάρχουν αυτοί οι ευρωπύραυλοι, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ακριβώς διότι ήταν ένα εργαλείο για να ε, αναγκάσουμε τη Σοβιετική Ένωση τότε να υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Ήταν πάρα πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε ένα έγγραφο της Στοκχόλμης μετά την υπογραφή της συνθήκης όπου πραγματικά υπήρχαν ομάδες ελεγκτών και από, τη, από τη μία πλευρά που πήγαινε και έκανε ελέγχους στην άλλη πλευρά σε πυράβλους, πυράβλους βαλιστικούς, πυράβλους κρούς κτλ. Αυτό επετεύχθη λοιπόν μέσα στην πρώτη δεκαετία ε, ε, ισχύως της συνθήκης υπήρξαν ε, οργανωμένες καταστροφές πυρηνικών κεφαλών οι οποίες είχαν συμφωνηθεί και υλοποιούνταν εκ παραλίλου και στις δύο πλευρές. Η Ειδική Επιτροπή Επαλήθευσης ε, ολοκλήρωσε το έργο της το 2001 μετά την ε, εκπνοή της φοιτείας ε, της στην 21η συνάντησή της συγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Όλα όσα είπα ε, μοιάζουν πολύ με την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Το νέο σύστημα πυράβλων του, της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ δημιουργούν ένα πολύ παρόμοιο σκηνικό όπως αυτό που δημιουργήθηκε με, το, με τους SS-20. Αποτελούν απειλή προς την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και, την, και, και ενισχύει τις δυσκολίες πυρηνικού ανεφοδιασμού. Έχει δημιουργεί, τα νέα συστήματα της Ρωσίας δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο ΝΑΤΟ όσον αφορά τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση. Ελπίζω αυτή η ιστορική αναδρομή να, σας, ε, να φώτισε λίγο το, πόσο σημαντική, για ποιο λόγο είναι σημαντική αυτή η συνθήκη ε, INF. Ακριβώς διότι ανάγκασε ε, της ήπα και την Σοβιετική Ένωση να αποφύγουν θερμό επεισόδιο πυρηνικό. Δεν ήταν απλά λόγια, πραγματικά εξασφάλισε η συνθήκη αυτή τη σταθερότητα που χρειαζόμασταν στο τέλος του ψυχρού πολέμου. Γι' αυτό ε, οι σύμμαχοι επιμένουν στη συνθήκη αυτή εξακολουθούν να καλούν τη Ρωσία να επανέλθει σε πλήρη συμμόρφωση. Είναι κρίσιμη σημασία ζήτημα για μας, για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, των συμμάχων και όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Διευθυντά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε για την ιστορία του ΝΑΤΟ. Ελπίζω να μπορούμε να έχουμε και γραπτά κάτι για να το μοιράσουμε στους ευρωβουλευτές μας. Ε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ωραία και πάλι καλώ ήρθατε κύριε Πάιφερ, ο πρέσβης. Θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ με τον Γιάτσεκ Μπιλίτσα και τον Βίλιαμ Αλμπέρκα. Εδώ είμαι ως εξωτερικός ε, συνεργάτης του Ιδρύματος Brookings, θα μιλήσω όμως εδώ προσωπικά και όχι εκ μέρους του. Και θα σας μιλήσω για το μέλλον κυρίως της συνθήκης INF μετά την περιγραφή που είχαμε. Και θα μιλήσω και για τις επιπτώσεις στην περίπτωση που καταρρεύσει η συνθήκη αυτή και τι βήματα μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει συμμόρφωση. Είχαμε πρώτα τη ρωσική παραβίαση όσον αφορά τις δοκιμές και την ανάπτυξη του περίφημου 9M729 πυράβλου κρούς εδάφους που ονομάζουν SSC8 οι Αμερικανοί. Το Δεκέμβριο που μας ε, πέρασε υπήρξε ένα δημόσιο public στο ε, Ίδρυμά μας ε, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για το πώς θα αντιδράσουν στην παραβίαση αυτή της Ρωσίας και το έγγραφο πολιτική έλεγε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ε, δεσμεύεται πάντα υπέρ τη συνθήκη αυτή, αλλά επίση λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εξετάσει την κατάσταση και θεωρεί ότι είναι απαράδεκτη όσον αφορά την συμμόρφωση αυτή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε συμμορφώνονται, συνθήκη όχι όμω η Ρωσία. Και γι' αυτό χρειάζεται μια αντίδραση και η πρώτη θα ήταν διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η παραβίαση χρησιμοποιώντας μια επιτροπή επαλήθευσης που δημιουργήθηκε από ό,τι έμαθα για να συζητώνται εκεί τέτοια θέματα συμμόρφωσης. Δηλαδή, το δεύτερο θα ήταν ε, στρατιωτική αντιμετώπιση πρώτα απ' όλα με έρευνα και ανάπτυξη προγραμμάτων για να εξεταστούν αυτές οι ε, θέσεις των ΗΠΑ και να ξέρετε ότι το Κογκρέσο ήδη σκέφτεται να εμποδίσει την ε, έγκριση των 58 εκατομμυρίων δολαρίων ακριβώς εξαιτίας αυτής της ε, παραβίασης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια συμμόρφωση και μόνο σε αυτήν την ε, περίπτωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τη συνθήκη αυτή. Και ο τρίτο πυλώνα θα ήταν οικονομικά μέτρα κατά τη Ρωσία, κυρώσει ε, δηλαδή, μεταξύ άλλων όμω και ε, ανάπτυξη και παραγωγή 9M729. Στη συνέχεια δεν είχαμε πρόοδο όσον αφορά την συμμόρφωση αυτή. Το Δεκέμβριο, 20 Δεκεμβρίου, συζητήθηκαν κυρώσεις με την περίπτωση της Ρωσίας και το γραφείο Νόβατορ, όπως επίσης και την υπηρεσία Titan Central, που μπήκανε σε κατάλογο κυρώσεων. Τώρα στη συνέχεια. Να ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, το ναυτικό τη είχε τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τέτοιε ε, κεφαλές σε υποβρύχια ήδη από τη δεκαετία του 90. Και ο ε, Ομπάμα αναζωγόνησε αυτήν την ε, υπόθεση. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σε ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε για την πυρηνική θέση, ότι το σκέφτονται οι Ηνωμένε Πολιτείε να επαναργοποιήσουν τι κεφαλέ αυτέ και ότι ίσως ξαναδούνε τη θέση του Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τα πυρηνικά. Τώρα κάποια σχόλια για την προσέγγιση των Ηνωμένων Πρώτα απ' όλα, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη διπλωματική και την οικονομική πτυχή της προσέγγισης αυτής και συμφωνώ επίσης ότι χρειάζονται μέτρα διότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αλλάξει και να συμμορφωθεί αν δεν ξέρει ότι έχει να πληρώσει ένα πολύ βαρύ τίμημα. Όμως δεν ξέρω κατά πόσο η απάντηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι πιο σοφή. Η... Αν ανέπτυσαν και πάλι ε, πυράβλους μέσω συλλογικού οι Ηνωμένες στην Ευρώπη, μόνο τότε θα άλλαζαν οι υπολογισμοί της Ρωσίας. Οι κρούς εδάφους στην Ευρώπη τη δεκαετία του 80, παρά την αντίθεση του κόσμου, παρόλα αυτά ήταν στοιχείο κλειδί, γιατί έκανε τους Ρώσους να αλλάξουν την δικιά τους τακτική και να δεχτούν την απαγόρευση. Όμως, βέβαια, πολλά ερωτήματα τίθενται. Πρώτα απ' όλα, η έρευνα και ανάπτυξη δεν είναι κάτι τόσο ακριβό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα σοβαρό πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγή πυράβλων μέσου βιλινικούς, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα κοστίσει εκατομμύρια δολάρια τώρα που ο προπολογισμό των ΗΠΑ πιέζεται φοβερά. Δεύτερον, η ρωσική παραβίαση είναι κάτι που γίνεται τώρα. Οι πύραυλοι τώρα αναπτύσσονται και η αμερικανική απάντηση μετά από έρευνα και ανάπτυξη δικών τους πυράβλων θα λάβει χώρα μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, 3, 5, 7. Αλλά το τρίτο είναι ότι τέτοιοι αμερικανικοί πύραυλοι θα ανασαχίσουν το Κρεμλίνο μόνο αν εγκατασταθούν σε ρωσικό έδαφος ή τέλο πάντων σε μια πολύ γείτονο χώρα ή την Νότια Κορέα ή την Ιαπωνία. Τη δεκαετία του 80 εγώ ήμουνα στο ΝΑΤΟ και συμμετείχα σε διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις δυνάμεις αυτούς πυράβλους μέσου βιλενικούς και καταφέραμε να έχουμε μια τέτοια ανάπτυξη. Κανείς όμως δεν θα ήθελε να ξαναμπούμε ε, στο ίδιο πείραμα, στην ίδια δυσκολία. Οπότε αναρωτιέμαι, αν γίνει κάτι τέτοιο θα ανησυχήσει τη Ρωσία και θα την κάνει να αλλάξει τακτική. Δεν νομίζω. Ούτε είμαι σίγουρος ότι οι νέοι πύραυλοι εκτόξευσης θα αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί δεν πρόκειται η Ρωσία να συμμορφωθεί, από την άλλη μεριά ε, κινδυνεύουν να αλλάξουν και άλλα πράγματα προς το χειρότερο. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια στρατιωτική απάντηση, όποια και αν είναι. Μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερα συμβατικά στην Ευρώπη. Κάποιους ε, πυράβλους συμβατικούς, το B1 και το B2 για παράδειγμα, ή περισσότερες, ε, περισσότερα πολεμικά στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα υπευρύχιο το οποίο έχει 154 πυράβλους πάνω του στη Νορβική θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα, για να δείξουμε στη Ρωσία ότι μπορούν να υπάρχουν πυρηνικέ ικανότητες που θα αναπτυχθούν κοντά τους και θα τους απειλούν. Πρέπει έτσι να πείσουμε το, την Μόσχα να επιστρέψει στην συνθήκη και να ξέρει από τι κινδυνεύει. Τέτοια πράγματα με τις υπάρχουσες ικανότητες θα ήταν πιο αποδεκτά και στο ΝΑΤΟ και θα είχαν πιο γρήγορα αποτελέσματα από ότι το να αναπτύξει πυράβλους μέσου βεληνικούς η Αμερική. Και ένα άλλο σχόλιο όσον αφορά την ανησυχία μου σε περίπτωση κατάρρευσης της συνθήκης. Ως Αμερικανός εκπλήσωμαι από την σιωπή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο το 9M729 δεν μπορεί να πλήξει την Αμερική. Εκτός αν το βάζανε στη, στη βόρεια Ρωσία, ίσως όπου ποτέ δεν έχουν εγκαταστήσει πυράβλους. Μόνο τότε ίσως να έφτανε στην Αλάσκα το 9M729. Οι Ρώσοι αναπτύσσουν αυτό τον πυραβλό για να πλήξουν την Ευρώπη και την Ασία. Και το ΜΕΝΑ το έχει κάνει κάποιες δηλώσεις αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τον όρο ρωσική παραβίαση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, αλλά πουθενά δεν φαίνεται ότι οι ψηλά ιστάμενοι Ευρωπαίοι ε, θέτουν το ζήτημα αυτό στον πρόεδρο Πούτιν. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ε, δεν το κάνουν εκτός ε, ΝΑΤΟ. Και είναι λάθος αυτό. Είναι σφάλμα. Γιατί αν καταρρεύσει η συνθήκη αυτή για τα πυρηνικά μέσου βεληνικούς, τότε η Ευρώπη κινδυνεύει περισσότερο. Οπότε η σιωπή αυτή στέλνει ένα πολύ κακό μήνυμα στη Μόσχα, δείχνει ότι η Ευρώπη δεν ανησυχεί γι' αυτό το συγκεκριμένο ε, πύραυλο, ούτε θεωρεί ότι παραβιάζει τη συνθήκη η Ρωσία. Χάνει δηλαδή η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χάνουν την ευκαιρία να πιέσουν περισσότερο διπλωματικά τη Ρωσία είναι λάθος. Τώρα πρόκειται για μια συνθήκη με τις Ηνωμένε Πολιτείε που δεν πάνε καλά οι σχέσεις Αμερικής και Ρωσίας. Είναι κάτι όμως που θα επηρεάσει Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Κορέα. Αλλά νομίζω ότι η σιωπή αυτή της Ευρώπης στέλνει ένα στραβό μήνυμα και προς την Ουάσιγκτον. Γιατί στην Ουάσιγκτον υπάρχουν κάποιοι στο Capitol Hill που πιστεύουν ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η Αμερική από τη συνθήκη αυτή, κάτι το οποίο θα ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου. Αλλά αν οι Ευρωπαίοι δεν διαμαρτυρηθούν για την παραβίαση της συνθήκη από πλευρά τη Ρωσία, δεν νομίζω ότι θα ακουστούν οι απόψεις τους για διατήρηση της συνθήκης από την Ουάσιγκτον. Φοβούμε λοιπόν ότι η συνθήκη αυτή πάει προς την κατέρευση, κάτι το οποίο θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των ΗΠΑ, της Ασίας και της ίδιας της Ρωσίας. Η Ρωσία, αν κατέρευσει τη συνθήκη αυτή, θα μπορούν να αναπτύξουν όσους 9 M729 θέλουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα μπορεί να αναζωογονήσει και τους SS20 αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα πλήξει πάρα πολύ την ασφάλεια σε Ευρώπη και Ασία. Το δε πεντάγωνο από τη δικιά του την πλευρά θα αρχίσει να αναπτύσσει τους δικούς του πυράβλους μέσου βεληνικούς. Οπότε θα τεθεί το ζήτημα και στην Ευρώπη τότε. Πάντω η κατάρρευση τη συνθήκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη συνθήκη αυτή καθευτεί. Πιστεύω ότι θα επηρεάσει και γενικότερα το καθεστώ ελέγχου των πυρηνικών ΗΠΑ Ρωσίας. Υπάρχει το New Start που στο Φεβρουάριο θα αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή, να υλοποιείται και τι θα γίνει εφόσον δεν συμμορφώνεται η Ρωσία. Το 2021 εκπνέει η συνθήκη και θα μπορούσε για πέντε χρόνια να παραταθεί χωρίς να χρειάζεται να πάει για επικύρωση στη Γερουσία. Πιστεύω ότι το New Start προσφέρει πάρα πολλά στην ασφάλεια Αμερικής, Ευρώπης και Ρωσίας. Αν όμως δεν υπάρχει η συνθήκη ΕΝΕΦ ή αν παραμένει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ρωσία συμμορφώνεται ή όχι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε το New Start να το παρατείνουμε. Ήδη σας είπα ότι το Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι κυρίως, προσπαθούν και το λένε να εμποδίσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν κονδύλια για παράταση του New Start, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η Ρωσία συμμορφώνεται στη συνθήκη για το πλεμέσου βεληνικούς. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν καταρρεύσει η συνθήκη και δεν ε, παραταθεί το New Start, θα είναι η πρώτη φορά για 45 χρόνια που δεν θα υπάρχει συμφωνία που να περιορίζει τα πυρηνικά στι ΗΠΑ και τη Ρωσία. Κάτι το οποίο θα έχει πολύ σημαντικέ συνέπειε. Πρώτα απ' όλα, αν δεν υπάρχει το New Start, δεν θα υπάρχει περιορισμό, δεν θα υπάρχει ούτε ανταλλαγή πληροφοριών, ούτε κοινοποίηση, ούτε επιθεωρήσει που έχουμε μέχρι τώρα και που προσφέρουν πάρα πολλέ πληροφορίε και που βέβαια θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα αλλιώς στις ΗΠΑ να τις αποκτήσουν. και θα χρειαστεί να γίνουν πολύ πιο ακριβές αποφάσεις να παρθούν όσον αφορά τον εξοπλισμό. Αν δεν υπάρχει το New Start, ούτε η Washington ούτε η Μόσχα περιμένω να αναπτύξουν πολύ περισσότερο το δυναμικό τους πέρα από το New Start, αλλά ποιος ξέρει, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα έχει λίγο κεφαλές η Ρωσία θέλει να αναπτύξει την ίδια ικανότητα και αν δεν υπάρχει περιορισμός γιατί να μην βάλει πολύ περισσότερες κεφαλές. Και όσον αφορά τις διμερείς πυρηνικές σχέσεις, τι θα γίνει με το καθεστώς μη διάδοσης πυρηνικών. Η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το 90% των πυρηνικών ε, του κόσμου ολόκληρου. Οπότε αν οι ίδιε δεν περιορίζουν τα πυρηνικά του, πώς θα πετήσουν από τρίτε χώρες να μην αναπτύξουν περισσότερο τα δικά τους πυρηνικά. Και ανησυχώ ιδιαίτερα για τις αντιδράσεις τη Κίνας. Η Κίνα τα τελευταία 25-30 χρόνια προσπαθεί να αναπτύξει πυρηνικά, βέβαια με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Όμω την έχουν πάρει την απόφασή του. Ξέροντα, αυτή να μην αναπτύξουν γρήγορα δηλαδή τα πυρηνικά, ξέροντα ότι υπάρχει ο περιορισμός στις ΗΠΑ και στη Ρωσία. Αν δεν υπάρχει πια αυτό, τι θα κάνει η Κίνα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ φοβάμαι ότι θα είμαστε σε έναν κόσμο λιγότερο σταθερό και λιγότερο ασφαλή σε αυτή την περίπτωση. Ελπίζω να σωθεί η συνθήκη INF και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Και θα μπορούσα να κάνω κάποια σχόλιο και μετά να απαντήσω ερωτήσεις για το τι βήματα μπορούν να γίνουν για να διατηρηθεί η συνθήκη αυτή. Η ίδια η Ρωσία κατηγορεί για τρία πράγματα για παραβιάσει στι ΗΠΑ τη συμφωνία αυτή. Υπάρχει τρόπο όμω να αντιμετωπιστούν αν υπάρχει καλή βούληση. Και ελπίζω να υπάρχει και να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρεσβευτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Έλερ. Παρακαλώ. κύριε Πρεσβευτά. Εκτιμώ αυτά που είπατε. Εγώ αναφέρθηκα στην υποκριτική στάση της Ένωσης. Σωστά είπατε ότι οι αρχηγοί κρατών δεν έχουν πει τίποτα τα τελευταία ένα-δυο χρόνια. Αν όμως το δείτε αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, Σημαίνει ότι έχουμε χάσει περίπου ένα χρόνο διαβεβαιώνοντα ο ένα τον άλλο ότι θα τηρήσουμε τι πολυμερεί συμφωνίε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είχαμε και μια χαμένη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, όπου είπαμε ότι εντάξει, θα παραμείνουμε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν φτάνει. Αν δείτε και τα πρακτικά που δημοσιεύονται προσεκτικά, δεν υπήρξε καμία αναφορά από την Αμερικανική πλευρά στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ για την συνθήκη αυτή. INF. Αλλά αυτό το θέμα δεν είναι νέο. Μας απασχολεί πολιτικά εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Οπότε αυτό το έτος χάθηκε και για τις δύο πλευρές. Είναι χαμένο. Εγώ στην πολιτική μου ζωή είδα ότι δεν ήταν project η παρουσία των Πέρσιν στην Ευρώπη. Δεν ήταν έτσι κάτι το πολύ δημοφιλές, αν κάποιος ήταν υπέρ της παραμονής τους ή της παρουσίας τους αλλά υπάρχει ένα αίσθημα απογοήτευσης και ένα ερωτηματικό. Γιατί αν οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις φαίνεται τελικά να είναι μία σχέση μεταξύ δύο μεγάλων ανδρών, πέρα από τις διμερείς συμφωνίες, τότε υπάρχει η εντύπωση ότι Οι ανησυχίες των ΗΠΑ δεν αφορούν τους συμμάχους τους, σε σχέση δηλαδή με την υποχρέωση που έχουν για να επιδείξουν βούληση για την τήρηση αυτών των πυράβλων στην Ευρώπη σε περίπτωση που αποσυρθούν από τη συνθήκη να φυρώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι λοιπόν να δεχτούμε αυτές τις αντιδράσεις γιατί για τις νέες χώρες της Ευρώπης εντάξει υπάρχει το θέμα των κυρώσεων προς τη Ρωσία το οποίο πλήττει την ανατολικογερμανική οικονομία. Δεν ξέρω κατά πόσο το πλαίσιο του ΝΑΤΟ έχει εδώ κάποιο ρόλο, αλλά είναι θέμα μεταξύ προέδρων, μεταξύ προσώμα, προσώπων που τα θεωρούν αυτά ως κατωτυπικό. Και πρέπει κανείς να δει ακριβώ την περιπλοκότητα και το περιεχόμενο αυτών των πολυμερών συμφωνιών. Γιατί φαίνεται να θεωρεί η κοινή γνώμη ότι θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ δύο ισχυρών ανδρών και ότι οι επιχειρηματίες και από τις δύο πλευρές θα ρυθμίσουν τα υπόλοιπα. Μπορεί να έχετε απόλυτα δίκιο ότι ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινή γνώμη πολιτικά και είναι αλήθεια ότι χάσαμε ένα έτος αφοσιωμένοι σε άλλα πράγματα, αστεία. Και οι Ρώσοι εξετάζουν ακριβώς την κοινή γνώμη στις χώρες του ΝΑΤΟ και χάσαμε χρόνο. Πρέπει πάντως να αντιδράσουμε και εγώ θα στείλω γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν ή στην κυρία Μογκερίνη γιατί πράγματι εμείς υποτιμήσαμε το γεγονός ότι εδώ έχουμε μία δημόσια συζήτηση στις χώρες της Βαλτικής, ακόμα και στην Πολωνία όπου θα ανέμενε κανείς κάποια ανησυχία για τις δράσεις της ε, Ρωσίας. Το θέμα αυτής της συνθήκης ΕΝΕΦ ποτέ δεν ε, αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση για το ότι θα κάνει βέβαια ο Πούτιν, εντάξει το αναφέρουν, αλλά όχι ακριβώς την δέσμευση των χωρών της Ευρώπης ε, σε σχέση με το τι σημαίνει στα σύνορά τους γιατί αφήσαμε την ε, διαμόρφωση της κοινή γνώμης σε ένα επίπεδο αφηρημένο όπου οι ισχυρές προσωπικότητες το πάλι θα βρουν λύσεις στα τέλος για όλα. Και παραμελήσαμε τελείως τη σημασία που έχουν αυτά τα περίπλοκα ζητήματα και οι μηχανισμοί περιπλοκών, περίπλοκων σχέσεων. Ευχαριστώ, ναι, Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε στην συνέχεια όσον αφορά την ε, πολιτική συνιστόσα και την συνθήκη αυτή. Ο κύριος Γκάλερ. Ο κύριε Λόζη. Μόλις ζήτησα το λόγο και σας ευχαριστώ που μου τον δίνετε. Πρώτο ερώτημα προς τον κύριο Πάιφερ. Παρακολούθησα τα όσα είπατε. Ωστόσο πρέπει να ομολογήσω ότι δεδομένου του 2017 υπήρχε η φήμη ότι υπήρχε ένα έγγραφο ε, εντός του ΝΑΤΟ για την εγκατάσταση που χαρακτήριζε την εγκατάσταση νέων πυράβλων ως μη ενδεδειγμένη λύση. Ε, παρατηρώ ότι... Εντάξει, μας είπατε βεβαίως τις δικές σας παρατηρήσεις, αλλά θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο εκτιμάτε ότι οι σχετικές σκέψεις στη ΣΥΠΑ έχουν προχωρήσει. Πόσο πιθανές δηλαδή θεωρείτε να, υπάρξει, πιθανό, θεωρείτε να, να έρευνα ε, αλλά και ανάπτυξη πυράβλων μέσω Στον κύριο Μπίλιτσα απευθύνω το εξής ερώτημα. Πολλές πλευρές ε, πολλές πλευρές ζητούν την εγκατάσταση νέων πυρηνικών κεφαλών στην Ευρώπη. Ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης αν πράγματι δηλαδή προχωρούσαμε σε εγκατάσταση ε, νέων πυρηνικών κεφαλών ε, στην Ευρώπη, όχι μόνο για τη συνθήκη INF, αλλά και για τις εν σχέσεις μας με τη Ρωσία. Και ένα ερώτημα προς τον κύριο Πάιφερ. Είπατε ότι το σημαντικότερο είναι να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και όχι μόνο να επαναλαμβάνουμε τι θέλουμε να κάνει η Ρωσία. Τι πιστεύετε εσείς λοιπόν ότι μπορεί να κάνουν η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασώσουν τη συνθήκη INF. Ποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για παράδειγμα θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι μπορούν να ληφθούν ε, ώστε να μην προχωρήσουμε, ώστε να μην υπάρξει κατάσταση ε, κλιμάκωσης. Για τον κύριο Αλμπέρκ. Εδώ και καιρό ε, κυκλοφορεί ένα έγγραφο αξιολόγησης ε, για τα μήνυ πυρηνικά όπλα. Εμφανίζεται πολύ συχνά στον τύπο το θέμα αυτό. Ακούγονται αυλαβείς, αυλαβεί αυτά τα μίνι ε, οπλικά πυρηνικά ε, συστήματα. Δείτε όμως τι έγινε στην ε, Χειροσύμα που με βάση τους όρους εκείνης της εποχής, μάλλον με βάση τους σημερινούς όρους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακριβώς ένα μίνι πυρηνικό όπλο. Ποια η θέση λοιπόν αυτών των μήνυ πυράβλων, των μήνυ πυρηνικών κεφαλών ε, στο πλαίσιο και των αμοιβαίων ελέγχων που γίνονται ε, βάσει της συνθήκης ε, INF και τι κίνδυνο θέτουν και δημιουργούν αυτές οι, αυτές οι μήνυ πυρηνικές κεφαλές για την ίδια τη συνθήκη INF. Ευχαριστώ κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους και για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ένα ερώτημα κατανόησης θέλω να σας θέσω. Ε, η συνθήκη για τους πυράβλους μέσου βελληνικούς συνήφθη πολύ πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την επανένωση των δύο Γερμανιών. Κατά την επανένωση των δύο Γερμανιών υπήρξε συμφωνία ότι το ΝΑΤΟ δεν θα ε, επεκταθεί προς Ανατολάς. Δυστυχώ αυτή η συμφωνία δεν είχε το χαρακτήρα συνθήκης, ήταν μια απλή συμφωνία λοιπόν. Αν όμως τώρα πια εγκαθιστούμε πυράβλους του ΝΑΤΟ πολύ ανατολικότερα από το σημείο στο οποίο βρίσκονταν ε, στο παρελθόν, δεν είναι λογικό να περιμένουμε μια αντίδραση της Ρωσίας. Το ερώτημα μου είναι, λοιπόν, είναι Μήπως δεν αρκεί να ασχολούμαστε μόνο με τους πυράβλους μέσου βελληνικούς. Μήπως θα έπρεπε να, να προβούμε σε μια πολύ συνολικότερη διαπραγμάτευση, να ξαναδούμε και να δημιουργήσουμε ενδεχομένως και μια νέα τάξη όσον αφορά τα πράγματα στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στη συνθήκη για, τα, για τους πυράβλους μέσου βελληνικούς. Ευχαριστώ κύριος Γκάλερ. Κύριε Μπούχνερ και η κυρία, η κυρία Λέζινγκ το ξέρει, γιατί ξέρει τι, τι ακριβώς βρίσκεται. Μπορείτε να φανταστείτε ότι στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν δηλαδή ε, γινόταν η πραγμάτευση της συνθήκης 2-4, ε, που ε, το, στα μέσα της δεκαετίας του 80, ε, όταν υπήρχε ακόμα το σύμφωνο της Μπορείτε να φανταστείτε ο Χέλμουτ Κόλ να πήγαινε στον Γκορμπατσόφ και να ε, έλεγε ότι οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, οι Τσέχοι, οι Τσεχοσλοβάκοι τότε ε, δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθούν στο Άτο. Μα δεν υπήρχε τέτοια προοπτική τότε. Έτσι κι αλλιώς. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην πιστεύετε και μην διακινείται αυτούς τους ε, μύθους. Ιστορικά κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο τότε. Ένας δυτικογερμανός καγκελάριος, όχι, δεν, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ούτε, ούτε δεν μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Κυρία Λέζ, η πρόεδρος, κυρία Λέζιν και κύριε Γκάλερ, είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε. Θα σας δώσω και την ευκαιρία να απαντήσετε ε, αργότερα. Αλλά τώρα έχει το λόγο ο συνάδελφος. Ακόμα και αν ε, μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει, προφανώς και δεν μπορούσε να συναυθεί μια τέτοια συνθήκη ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση που θα αφορούσε την Πολωνία, την Τσεχία και την Ουγγαρία. Θέλω να πω ότι ε, πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας ποιες είναι οι πραγματικότητες ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Και το πραγματικό δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ρωσία παραβιάζει τη συνθήκη. Βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι στην, ε, ε στη ΣΥΠΑ οι, οποίες, ε, οι οποίοι έχουν ε, κάθε συμφέρον να μην υπάρξει παράταση χρονική αυτής της συνθήκης. Αλλά αυτή αυτό δεν είναι κάτι που έχει σχέση με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και εκεί αναφερόταν και, η δήλωσή μου ε, που αφορούσε την παραβίαση της συνθήκης από την Ρωσία. Η κυρία Λόζιν. Τότε κύριε Γκάλερ να σας απευθύνω το εξής ερώτημα. Αυτό που έχω ακούσει πολύ συχνά από εσάς ε, θα ήθελα να, να το τεκμηριώσετε ιστορικά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας φέρω αποδεκτικό στοιχείο. Η πρόεδρος, κύριε Γκάλερ, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Αν θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι το οποίο δεν συνέβη, που απλώς δεν συνέβη. Πώς αλλιώς να το πω. Εσείς ισχυρίζεστε ότι συνέβη κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Και καθώς δεν είναι αλήθεια δεν μπορώ και να αποδείξω το ότι δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει λέει η πρόεδρο για να μην υπάρξει μια ενδογερμανική συζήτηση σε, αυτό το θέμα, σε αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και ύψιστης τη σημασίας, θα ήθελα να μην υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ σας αυτή τη στιγμή. Ε, ό,τι και να ε, ε, όποια άποψη και να έχει κανείς, αυτή τη στιγμή η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, οι βαλτικές χώρες είναι αξιόπιστοι εταίροι και μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στη συλλογική ασφάλεια και άμυνα. Και εγώ δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να συζητούμε για φορείς εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που μάλιστα προσπαθούν να υπονομεύσουν και να υποσκάψουν τη θέση του ΝΑΤΟ και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιστορία ε, γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε βεβαίως να επανεξετάσουμε και ζητήματα που αφορούν την καγκελαρία Κόλ, ε, ζητήματα που αφορούν ε, την περίοδο, των, ε, την περίοδο του 1980. Ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση στον κόσμο. Σας παρακαλώ λοιπόν να σταματήσετε αυτό το διάλογο. Όσον αφορά την ενότητά μας απέναντι στη Ρωσία, εγώ πιστεύω ότι οι κυρώσεις, ναι, προκάλεσαν κάποιες συζητήσεις, ιδίως στις νέες χώρες. Αλλά έχουμε και μια κουλτούρα, ξέρετε, ε, να υλοποιούμε τα αναγκαία βήματα προκειμένου να εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητά μας έναντι των εταίρων μας. Και η Πολωνία ε, ήταν πάντοτε ε, στην, ε, στην πρωτοπορία εκείνων που υποστήριζαν τις κυρώσεις. Να ακούσουμε τους ομιλητές μας. Κύριος Μπιλίτσα. specific... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση για την επανατοποθέτηση νέων πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη. Νομίζω ότι όλοι βέβαια Είμαστε ικανοποιημένοι, χαιρόμαστε για αυτά που συνέβησαν από τη δεκαετία του 80 με τεράστιες μειώσεις στους αριθμούς των πυρηνικών κεφαλών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τινούμε να ξεχνάμε και ίσως εδώ ο Βίλιαμ να μας δώσει πιο ακριβή στοιχεία ότι δεν υπήρχαν εκατοντάδες ή χιλιάδες αλλά δεκάδες χιλιάδες πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη ακόμα και σε χαμηλό τακτικό επίπεδο σε επίπεδο πυροβολικού, ναρκών κλπ. Είναι απίστευτο το πόσο πιο ασφαλείς έχουμε γίνει με αυτές τις συνθήκες όπως την INF και να μην αναφέρω κι άλλες κιόλας όπως το PNIS δηλαδή την πρωτοβουλία την προεκή πρωτοβουλία για τα τακτικά πυρηνικά όπλα τα οποία αποσύρθηκαν από κεντρικές αποθήκες. Δεν νομίζω λοιπόν κανείς να χαρεί με το ενδεχόμενο ή την προοπτική κατάρρευση αυτών των συμφωνιών και η Ευρώπη να επιστρέψει στο χείλος καταστάσεων ψυχρού πολέμου. Είχαμε και την κρίση στην Κούβα, την πυρηνική, για τα πυρηνικά θυμάστε με τους πυράβλους, Βερολίνο κτλ. Είχαμε επίσης κοινωνικοπολιτικές εντάσεις επίσης που ανέφεραν οι συνάδελφες στις εισηγήσεις τους τη δεκαετία του 70 και του 80, όπου είχαμε τοποθέτηση πυράβλων Pershing 2 στην Ευρώπη. Θυμηθείτε ότι κατέρευσαν κυβερνήσεις λόγω αυτού του γεγονότος. Στη Γερμανία είχαμε διαδηλώσεις με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στο δρόμο που διαμαρτυρόταν για την τοποθέτηση αυτών των ενόπλων. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είμαστε πραγματικά ευλογημένοι με αυτή την ιστορική εξέλιξη. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τα διαφυλάξουμε όλα αυτά. Και νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή ακριβώς εδώ η συζήτηση και το μήνυμα από το Κοινοβούλιο για τη διατήρηση αυτών των κεκτημένων. Βεβαίως υπάρχουν προ, προκλήσεις όσον αφορά αυτές τις συνθήκες για τον έλεγχο διάδοσης και τον περιορισμό των όπλων που στηρίζει η Ευρώπη. Αλλά και εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πριν από λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε μια νέα πρωτοβουλία στο Παρίσι για τη χρήση χημικών όπλων συγκεκριμένα. Η συνθήκη λοιπόν για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων παρουσιάζει βεβαίως κάποιες προκλήσεις, αλλά εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε και δουλεύουμε σκληρά για να πετύχουμε και το συνολικό μήνυμα το οποίο προέρχεται από τα ευρωπαϊκά όργανα και από το Κοινοβούλιο είναι η ενίσχυση και διατήρηση αυτού του συστήματος. που διαφυλάσσει αυτό το χοψιανό δόγμα ελευθερίας για όλους. Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής λοιπόν. Προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Βεβαίως εκεί όπου χρειάζεται αμυνόμαστε και ενισχύουμε την άμυνα, αλλά ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί το τωρινό πολύ χαμηλό επίπεδο πυρηνικών όπλων και ενδεχομένω θα μειωθεί περαιτέρω στην Ευρώπη. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλμπερκ. Ευχαριστώ πολύ. υπόθηκε ότι χάσαμε χρόνο. Αλλά να δούμε γιατί παραβιάζεται συνθήκη η Ρωσία. Αν δείτε τις αμερικανικές προσπάθειες το 2014 για την επίλυση του συστήματος αυτός, αυτού είχαν γίνει διμερός και δεν οδήγησαν πουθενά. Το 2016 επιτέλους ζήτησε, ζήτησαν, είπαν να ενεργοποιηθεί ο κατάλληλος μηχανισμός. Νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν λυθεί πολύ ήρεμα, πολύ απλά επειδή μέχρι τώρα αρνούνται την ύπαρξη αυτών των πυράβλων οι Ρώσοι και μόλις πρόσφατα το Δεκέμβριο αναγνώρισαν την ύπαρξή τους. Θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει λοιπόν το 2014. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ελέγχους γιατί ήταν τεχνικά εμφανές ότι υπήρξε παραβίαση της συνθήκης. Χρησιμοποιούσαμε λοιπόν τους μηχανισμούς της συνθήκης μέσω ΝΑΤΟ, μέσω Ένωσης και τα λοιπά, ώστε να τραβήξουμε την προσοχή των Ρώσων σε αυτά τα θέματα. Αλλά να είχαμε και την Ουκρανική κρίση. Και είδαμε ότι οι Ρώσοι αντιτάχθηκαν στην επέκταση της σφαίρας επιρροής της Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όπως είπε και ο Στίβ, τα συστήματά μας αφορούν ευρωπαϊκές και ασιατικές εγκαταστάσεις. Γιατί όμως αυτό είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που θεωρούσαμε ότι θα ήταν ο κόσμος πριν κάποια χρόνια, ο οποίος έχει αλλάξει. Για τις ενδεχόμενε επιλογές και τι έπεται. Νομίζω ξεκάθαρα είπα προσπάσαν να διαπραγματευτούν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Υπήρξε στήριξη από την Ένωση και τους συμμάχους και η εξέταση του ενδεχομένου στρατιωτικής απάντησης αλλά κατά πόσο αυτό θα είναι επιτυχές δεν ξέρω και δεν ξέρω κατά πόσο οι Ρώσοι βεβαίως έχουν διάθεση να εμπλακούν σε συζητήσεις για περιορισμό αυτών των όπλων. Και αν δεν υπάρχει σαφήνεια εκ μέρους της Ένωσης, τότε θα προχωρήσουμε. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε στη Ρωσία ότι δεν μπορούν να παραβιάζουν τις υποχρεώσεις ή να παραβλέπουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι προς αμοιβαίο συμφέρον η τήρηση αυτών των συνθήκων. Και θα πρέπει μέσω ελέγχων να δείξουμε στη Ρωσία ότι υπάρχουν και επιπτώσεις. Για τη Γερμανία με χώρες όπως η πρώην Σουσουδού και η Ρωσία. Τα πάντα πρέπει να είναι γραπτά. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε προφορικό επίπεδο. Τι διαστάσει έχουν και οι Ρώσοι. Μια χειραψία δεν φτάνει. Δεν είναι αξιόπιστη. Οι Ρώσοι βέβαια δεν εμπιστευόταν αυτούς τους αναγκαλισμούς με τη Δύση. Πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας σοβαρά ως αντιπάλους. Δεν θα είναι συνεργάσιμος και αξιόπιστος σύμμαχος ή εταίρος. Περισσότερο ήδη θεωρούν τον εαυτό τους ως ανταγωνιστή μας. και κατά τη διάρκεια της καριέρας μου ασχολήθηκε με ένα πρόγραμμα που καθιστά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ρωσικές ασφαλής. Νομίζω πάντως ότι υπάρχει τρόπος να πείσουμε τους Ρώσους να έχουν άλλη στάση υπέρ της δικής ασφαλείας. Επίσης, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε, πρεσβευτή Πάιθερ. Ένα σχόλιο για το γερμανικό ζήτημα και μετά για την μη διάδοση. Τι διασφαλίσεις δόθηκαν στη Ρωσία στην επανένωση της Γερμανίας. Αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί πολύ. Εγώ έχω τη δικιά μου άποψη γιατί το 1998 ήμουνα στο Υπουργείο Εξωτερικών αρμόδιος για το θέμα αυτό με τη Ρωσία και είχαν γίνει συνομιλίες ε, με τον Υπουργό Μπέικερ και τον Σεβανάτζε και είχαμε περιοριστεί ότι δεν θα υπήρχαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην τέως Ανατολική Γερμανία. Εγώ έτσι θυμάμαι τις συζητήσεις. Ο κόσμος τότε δεν ε, σκεφτόταν όλα αυτά για το σύμφωνο της Βαρσοβίας κλπ. Για το θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών. Το 2017 δεν ήταν ότι καλύτερο, αλλά υπάρχουν και λόγια να το κατανοήσουμε ότι η κυβέρνηση χρειαζόταν χρόνο να εξετάσει τα ζητήματα, να καταλήξει στη δική της πολιτική. Και η κατάσταση όμως το Δεκέμβρη ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Και πολλοί ε, λένε στην κυβέρνηση ότι όντω η Ρωσία παραβιάζει τη συνθήκη. Και εγώ δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Ότι αναπτύσσουν τους πυράβλους του η Ρωσία προφανώς και το κάνει. Όχι όμως όχι όμως συνολικά. Τους πήρε χρόνο να καταλήξουν εκεί που καταλήξαν, αλλά ήταν καλό. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι η απόφαση των ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο, ήταν να γίνουν έρευνες και ανάπτυξη για τα συμβατικά μέσω Ε, εντάξει, μεν, αλλά το Δεκέμβριο μιλούσαμε για τα πυρηνικά και για το πόσο έχει προχωρήσει το πρόγραμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αλλά είμαι εκτό τώρα, έτσι, οπότε δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρω καλά. Τους τελευταίους 6-12 μήνες συζητάμε για την έρευνα και την ανάπτυξη πυράβλων μέσου βεληνικούς και με τους ε, στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών ε, παλιότερα ήταν περισσότερο θέμα και όχι τόσο Ευρώπης. Πιο πολίτη θα κάνουν με την Κίνα. Στην άλλη ερώτηση για το τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για να αλλάξει η κατάσταση, η απάντηση μου είναι εξή. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και η Ευρώπη πιστεύω ότι πρέπει να κάνει περισσότερα, να ασκήσει μεγαλύτερη διπλωματική πίεση στη Ρωσία. Θα ήταν καλό να έχουμε μια κατάσταση όπου ο Πούτιν ακούει και από την Ευρώπη. Κάθε φορά που μιλάμε με τους Γερμανούς, τους Ούγκρους, τους Πολωνούς, τους Ταλούς, τους Ιάπωνες ε, κλπ. Να τους λένε γιατί εσείς ε, στοχεύετε τη χώρα μου, γιατί βάζετε αυτούς τους πυράβλους που κινδυνεύουν να πλήξουν τη χώρα μου. Να το λένε ξανά και ξανά. Και σας είπα ότι οι πυράβλοι αυτοί δεν πρόκειται να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει περισσότερο θέμα με την Ευρώπη παρά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε η πολιτική πίεση πρέπει να γίνει απέναντι στους Ρώσους. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν στρατιωτικά αντίμετρα αξιόπιστα. Και εδώ είναι που ανησυχώ, γιατί θεωρώ ότι η απάντηση των ΗΠΑ δεν είναι στο ύψο που θα έπρεπε. Η αξιοπιστία της αμερικανικής απάντηση καταλήγει στο ότι η Ρωσία δεν ε, θα πληγεί από τίποτα. Και δεν ξέρω εσείς ε, τι λέτε, αλλά το 98 το θυμάμαι. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν αντιδράσει. Και ο πρέσβης ε, Νίτσε πίστευε ότι δεν θα γίνει η ανάπτυξη τότε. Γι' αυτό και δεν έλαβε υπόψη του τις διαπραγματεύσεις και πήγε βόλτα με τον ε, Ρώσο ομόλογό του για να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συμφωνία. Έκανε λάθος τότε. Γι' αυτό όμως και άλλαξε η ρωσική προσέγγιση, γιατί αναπτύχθηκαν τα συστήματα τότε. Τώρα δεν τον έχουμε, τον Σεβαρνάτσε, τώρα έχουμε τον Πούτιν. Και δεν θέλουμε βέβαια να μπούμε σε μια συζήτηση Αμερικής Ευρώπης για την ανάπτυξη των πυράβλων. Τη δεκαετία του 80 οι Ρώσοι προσπαθούσαν να κερδίσουν την κοινή γνώμη κατά της εγκατάστασης των πυράβλων αυτών. Τώρα πάλι η Ρωσία με τα κοινωνικά μέσα και τον χώρο θα έκανε ό,τι μπορούσε για να παρέμβει σε αυτή τη συζήτηση. Και δεν θα έπρεπε. Και το τρίτο που έχει να κάνει με την Αμερική είναι ότι οι Ρώσοι έχουν κατηγορήσει για τρία πράγματα την Αμερική, ότι παραβιάζει τη συμφωνία. Τα δύο εύκολα λύνονται. Αλλά υπάρχουν και ένα τρίτο όπου καταλαβαίνω τι εννοεί η Ρωσία όταν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση. Ε, πρόκειται για την περίπτωση της ε, Ρουμανίας και της ε, Πολωνίας για τις δοκιμές που γίνονται με τέτοιους πυράβλους. Πρόκειται για ένα σύστημα που υπάρχει σε αμερικανικά πλοία και μπορεί να μην έχει μόνο ένα SM3 αλλά και πυράβλους κρούς που θυμίζουν πάρα πολύ εκείνους εδάφους που περιλαμβάνει η συνθήκη. Και οι Ρώσοι λένε εμείς που ξέρουμε ότι δεν έχετε και πύραυλο κρούς. Αυτό θα μπορούσε κάπως να λυθεί για να μην ανησυχεί η Ρωσία. Αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να ε, βρει τρόπους να μας καθισκάσει όσον αφορά τον 9M729, ε, τότε και η Αμερική θα μπορούσε να πει εντάξει, τότε και εμείς ελάτε να ελέγξετε και να δούμε. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση αν αρχίζαμε από τον 9M729. Ευχαριστώ. κύριος πάλι και μετά θα πάρω και εγώ το λόγο. Νομίζω ότι καταλάβαμε το μήνυμα. Εσείς αναφέρεστε στα μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης. Και ορθώς. Αν μου επιτρέπετε όμως, θα ήθελα να πω ότι οι ΙΠΑ προσπαθούν με ήπιο τρόπο να προωθήσουν τις θέσεις τους μέσω διπλωματικών οδών κτλ. Παρά, όλα αυτά, δεν πρέπει κανείς να υποτιμά το γεγονός ότι η ρητορική που έχει αναπτυχθεί ιδίω στο Twitter υπονομεύει την προσέγγιση που έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε. Στη Γερμανία, μάλιστα, ε, έχουν, έχει πέσει και κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Και είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς πολιτικούς κύκλους. Μην υποτιμάτε λοιπόν τη σημασία που έχει το θέμα. Τα, αν ανατολικά κράτη που συμμετέχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν μια πιο ρεαλιστική άποψη για τη Ρωσία βοήθησαν στο να δημιουργηθεί μια εικόνα και στα άλλα κράτη-μέλη, στα παλιά κράτη-μέλη. Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 80 λόγω της Ένωσης και λόγω της αντίληψης που ε, έχει εγκατασταθεί στην κοινή γνώμη και στα άλλα κράτη-μέλη και στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι οι ΙΠΑ εξακολουθούν να είναι η φωνή του ελεύθερου κόσμου. Και παρόλο που αυτό μπορεί να έχει μια συμβολική αξία, αν δείτε τον γενικό πληθυσμό, η σημασιολογία και ο συμβολισμός αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις αντιλήψεις που υπάρχουν στον κόσμο. Όταν λοιπόν χειριζόμαστε ζητήματα όπως είναι η πυρηνική ισχύς με όρους εγώ το έχω μεγαλύτερο το κουμπί, τότε καταλαβαίνετε ότι υπονομεύεται και υποσκάπτεται η ασφάλεια. Γιατί βλέπετε ότι η κοινή γνώμη μπορεί όταν το επίπεδο έχει πέσει τόσο χαμηλά να επηρεαστεί πολύ εύκολα και από τη ρωσική προπαγάνδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό και θα πρέπει να σκιαγραφεί το πρόβλημα αυτό ως ευρωπαϊκό μεν, αλλά καλό θα ήταν ε, να μπορεί και ο κάθε πολίτης να μπορεί, να μπορεί ο κάθε πολίτης να ταυτίζεται με τη στάση που θέλουμε να διαμορφώσουμε εμείς απέναντι ε, στο πρόβλημα με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Νομίζω, λέει η Πρόεδρος, ότι η σημερινή συζήτηση μας βοήθησε να κατανοήσουμε τα ζητήματα με πιο ολοκληρωμένο και σφαιρικό τρόπο. Έχουμε σχηματίσει μια πιο σφαιρική άποψη για τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Η δική μου οπτική, όχι μόνο ως Ευρωβουλευτή, αλλά και ως εκπρόσωπο της περιοχής μας, ε, είναι ότι οι διατελετικές σχέσεις αποτελούν τον πυρήνα της ασφάλειας μας. Αυτό βεβαίως δεν αποκλεί, το αντίθετο μάλιστα, συμβαδίζει με την αναγνώριση από πλευράς μου του θετικού αντικτύπου που είχε στην πολωνική κοινωνία και σε άλλες κοινωνίες η προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από άποψη ασφαλείας όχι μόνο από άποψη ευημερία, δηλαδή που προσέφερε η προσχώρηση αυτή στους λαούς μας. Ταυτόχρονα, εγώ συμμετείχα στην ε, πολωνική αντιπολίτευση επί ε, κομμουνιστικού καθεστώτος και θυμάμαι πάρα πολύ καλά την περίοδο εκείνη και πρέπει να σας πω ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ακόμη και να υποφέρουμε προκειμένου να δείξουμε στην Ρωσία ότι ήμασταν ζωντανοί και για να τις, ασκήσουμε, για να τις ασκούμε πίεση. Βεβαίως οι εποχές αλλάζουν και το ίδιο ισχύει και για την ε, ε, ρωσική πολιτική και έπειτα από μια περίοδο ε, ομφαλοσκόπησης φαίνεται ότι εμφανίζονται με μεγαλύτερη ε, έμφαση πια οι ρωσικές φιλοδοξίες για ε, άσκηση επιρροής και ακόμη περισσότερο σε χώρες που δεν συμμετέχουν ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν για παράδειγμα. Γνωρίζω ωστόσο επίσης ότι όταν ξεκίνησαν συνομιλίες Ρίγκαν Γκορμπατσόφ η, των, των συζητήσεων αυτών είχαν προηγηθεί ε, μακροχρόνιες εργασίες ομάδων εμπειρογνωμόνων και από τις δύο πλευρές. Δεν ήταν λοιπόν μόνο προσωπικό το θέμα μεταξύ της χημίας Ρίγκαν και Κορμπατσόφ, υπήρχε μια ολόκληρη προεργασία Εγώ λοιπόν προσωπικά κιόλα, ενδιαφέρομαι πάρα πολύ όχι μόνο ε, για την ε, αξιολόγηση προσωπικών χαρακτηριστικών αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ε, σχηματίζουμε μια πολύ συνολικότερη εικόνα. Ναι, συμφωνώ, πρέπει να ενισχύσουμε τη διπλωματική πίεση που ασκούμε αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές κατά την αξιολόγηση όλων των παραγόντων. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, προτιμώ οι ΙΠΑ να είναι ισχυρές. Αυτά είχα να δηλώσω εγώ. Αν δεν έχουν κάτι άλλο να προσθέσουν και οι προσκεκλημένοι μας, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και τους τρεις για, την για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Τα μέλη της Επιτροπής βεβαίως για τη συζήτηση. Και παρότι δεν ήμασταν τόσο πολύ όσο στο προηγούμενο θέμα, θεωρώ ότι το θέμα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολλά ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας θα γίνει στις 26 και 27 Φεβρουαρίου. Διήμερη συνεδρίαση και πάλι. Υπάρχει κάποιο θέμα στα διάφορα που θα θέλετε να συζητήσουμε. Όχι ούτε παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και ως συνήθως βεβαίως και τους διερμηνείς μας για το εξαιρετικό τους έργο. Σας ευχαριστώ και γεια σας.